Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και σας ευχαριστώ θερμά. Να σας ζητήσω συγγνώμη καταρχήν για μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Γιατί δεδομένη τη ε, συνέχισή των συζητήσεων μεταξύ εισηγητού και σχεδόν εισηγητών, αλλά και τη συζήτηση πολιτικέ πολιτικές ομάδες και τη δυνατότητα να ε, εκπονηθούν κάποιε συμβαστικέ τροπολογίε για να καλύψουν την πληθώρα των άλλων τροπολογιών. Υπάρχει πρόταση και έγινε δεκτή για αναβολή της ψηφοφορίας τη έκθεσης του κυρίου Αντριέ ε, που θέμα έχει του τρόπου με του οποίου μπορεί η κοινή γεωρική πολιτική να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ήπεθρο. Πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα. Και, και σίγουρα ε, θα εμπλουτιστεί από τα πορίσματα της διάσκεψης που έγινε Δευτέρα και Τρίτη ε, και που επανέλαβε ε, μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει το 1996 ε, μετά από πρωτοβουλία του Επιτρόπου Φίσλερ και μετά από μια σημαντική διακήρυξη που έγινε τότε. Πολύ σημαντική και αυτή η διάσκεψη που έγινε τώρα στο ΚΟΡΚ. Χάρη στη διακήρυξη εκείνη, η διακήρυξη οι διατάξεις ε, ε, της μεταγενέστερης μεταρρύθμισης της ε, ΚΑΠ έλαβαν υπόψη και την ανάπτυξη στην Ήπεθρο και την ε, δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης εκεί. Και μάλιστα η, διάσκεψη της 5ης και 6ης ε, Σεπτεμβρίου στο ΚΟΡΚ ακριβώς συνέχισε την προηγούμενη ε, διάσκεψη και πραγματεύτηκε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πέθρος ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και μάλιστα συμμετείχε και ο κύριος Φίσλερ που ήταν ο πρωτεργάτης της πρωτοβουλίας αυτής πριν από 20 χρόνια. Είναι σκόπιμο λοιπόν να ενημερωθούμε και εμείς για τα αποτελέσματα αυτής της συνδιάσκεψης του ΚΟΡΚ και να τα λάβουμε υπόψη στην περαιτέρω διαμόρφωση των εργασιών μας, αλλά και την εκπόνηση της έκδοσης του κ. Αντρία. Ε, στην ε, διάσκεψη αυτή έλαβαν μέρος και ο Επιτροπός Φίσλερ, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εκπρόσωποι του ΩΣΑ, Υπουργοί Γεωργίας, της Σλοβακίας ε, που ασκεί την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν πολύ σημαντική, όπως είπα, η διάσκεψη. Οπότε, το σημείο αυτό αναβάλλεται, το σημείο 3. Έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες με εξαίρεση στονικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και γορδελικά. Η μέρη σε διάταξη εγκρίνεται. Και να περάσουμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, την έκθεση του κυρίου ΕΚ. Παρακαλώ κύριε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω δύο ε, παρατηρήσει για την σε διάταξη και επειδή συνήθω εργάζεται σοβαρά η Επιτροπή μα, πρέπει να πω ότι λάβαμε ένα έγγραφο, μια έκθεση που δεν βρίσκεται καθόλου στο πνεύμα του Κοινοβουλίου. Το πρωτότυπο είναι στα πολωνικά. Αλλά εδώ μα έχει έρθει στα χέρια ένα έγγραφο στα αγγλικά. Ε, δεν είναι έτοιμε μεταφράσει και το πρέπει να το έχουμε μελετήσει. Ε, δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό. Σα παρακαλώ λοιπόν, Πρόεδρε, όταν ετοιμάζετε μια έκθεση να φροντίζετε να ε, μπορούν όλοι να έχουν κατανόηση του κειμένου. Έπειτα. Δεν ξέρω γιατί καλέσαμε τη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας σήμερα. Αλλά είναι πολύ στενή ημερή σε διαταξή πέρα από την προστασία των ε, προς εκτροφή κουνελιών. Πιστεύετε, Πρόεδρε, ότι το πιο σημαντικό θέμα είναι η έκταση των περιφραγμάτων και το αν τα κουνέλια είναι ευτυχισμένα σε συνθήκες εχμαλωσίας. Νομίζω ότι έχουμε πολύ σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε, όπω οι καταστροφικέ οδιέ των Δημητριακών αυτό το καλοκαίρι. Οι γεωργοί μα σήμερα έχουν σοβαρότερε δυσχέρειε. Ε, και πολλέ φορέ ε, δεν μπορούν να ζήσουν την οικογένειά του. Ε, εδώ λοιπόν, Πρόεδρε, θέλω να το επισημάνω αυτό, διότι αν το θέμα σα είναι απλώς να είμαστε αρεστοί στο κοινό και να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο, ε, δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό. Έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε στην Επιτροπή μας. <clears throat> Ε, εύστοχη παρατήρηση για τη μετάφραση. Θα γίνει μετάφραση στα γαλλικά. Και η επιλογή των πολωνικών εξηγείται από το γεγονός ότι ήταν δική μου η πρωτοβουλία. Και προσπάθησα να το επισημάνω στον εισηγητή και τελικά ε, κατάθεσα και δική μου πρωτοβουλία για τις ε, εξωτερικές πτυχές, τις πτυχές εξωτερικής πολιτικής και πόσο επηρεάζουν την κοινή γεωργική πολιτική και την κατάσταση των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι έχει νόημα να κάνουμε μια ευρυθή ανάλυση της εξωτερικής αυτής διάστασης και πώς επηρεάζει αυτή την κοινή γεωργική πολιτική. Επίσης να λεφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη γεωργία. Γιατί πολύ συχνά έχουμε την εντύπωση ότι η γεωργία παραμελείται ή χρησιμοποιείται μόνο για την ε, ε, ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών. Επίσης, ε, έχουμε πολλές επιμέρους αγορές και πολύ συχνά ασχολούμαστε με την κατάσταση στις γεωργικές αγορές. Και αυτή τη στιγμή κάνουμε ανάλυση γενικώ της ε, κατάστασης στην αγορά των Δημητριακών, γιατί όντω και εκεί υπάρχει κρίση και έχουμε και τεράστιες εισαγωγέ ε, Δημητριακών από την Ουκρανία αλλά και από άλλε περιοχέ του κόσμου. Οπότε σίγουρα θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό γιατί όντω είναι πολύ σημαντικό. Οπότε θα ήθελα να παρουσιάσετε και στην ε, δική σας πολιτική ομάδα αυτή την πρωτοβουλία και να συνεννοηθούμε μετά στους συντονιστές πότε θα τη δρομολογήσουμε ε, και στην Επιτροπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των κουνελιών, εδώ και καιρό ασχολούμαστε με το θέμα αυτό των εκτρεφόμενων κουνελιών που έχει και οικονομική διάσταση αλλά και διάσταση ε, ευζωίας καλής μεταχείρισης των ζώων. Γι' αυτό και το θέσαμε και πάλι στην ημερήσια διάταξη. Γιατί και το θέμα των κουρελιών είναι σημαντικό. Οπότε περιμένουμε την ε, παρουσίαση της έκθεσης του κύριου Εκ που θα μας πει ακριβώς για τη σπουδαιότητα του θέματος. Η πρώτη παρουσίαση έχει γίνει τον Ιούνιο, 21 Ιουνίου παρουσίαση του εγγράφου εργασία. Σήμερα θα γίνει παρουσίαση του σχεδίου έκθεση. Οπότε μπορώ να δώσω το λόγο στον εισηγητή μα τώρα, στον κύριο Εκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εκπρόσωποι της Κομισιόν και του Συμβουλίου, Αξιότιμο κύριε Πρόεδρε. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την έκθεση πρωτοβουλίας, μας, μου για τους στοιχειώδες κανόνες εκτροφής των κουνελιών. Όπως γνωρίζετε, ο αριθμός των λέξεων για την ε, σύνταξη μιας έκθεσης είναι περιορισμένος. Γι' αυτό το λόγο επικεντρώνομαι στην καταλληλότητα για την τήρηση και την εκτροφή κουνελιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοώ τις ε, κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις του θέματος. Και σε κάθε περίπτωση θα λάβω υπόψη μου και τις δικές σας προτάσεις. Πριν από το καλοκαίρι σας παρουσίασα το έγγραφο εργασίας μου και σας είπα ότι με αυτή την έκθεση επιδιώκω πολλαπλούς στόχους. Πρώτον, ο κύριος στόχος για μένα είναι να κλείσουμε το κενό στην ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς δεν υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των κουνελιών ε, στη Γεωργία. Δεύτερον, ως μεσοπρόθεσμο στόχο έθεσα ε, το να δοθεί στον κλάδο η δυνατότητα να ε, αξιοποιήσει μεθόδους παραγωγής με επίκεντρο τον καταναλωτή προκειμένου να μπορέσουν να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά. Και τρίτον, ως φραχυπρόθεσμο στόχο ε, έθεσα να ξεκινήσει η συζήτηση για την εμπορική εκτροφή κουνελιών. Μία ε, αναφορά με περισσότερες από 6.000 υπογραφές ε, των Ευρωπαίων πολιτών με απεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν και την, ε, ε τους Υπουργούς Γεωργίες είναι απόδειξη για το γεγονός ότι το δημόσιο ενδιαφέρον αυξάνεται για αυτό το θέμα. Επίσης, η συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους στη διάρκεια του καλοκαιριού μου έδειξε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν κοιτάξει κανείς τα κονικλοτροφία στην Ευρώπη, θα δει ότι ο κλάδος αυτός βρίσκεται σε φθήνουσα πορεία. Τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαρκώς διαπίστωσαν μια μείωση της παραγωγής τους και οι προβλέψεις για το έτος 2016 δείχνουν ότι θα έχουμε μια μείωση της τάξης του 4%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σαφής τάση και έτσι και τα επόμενα χρόνια η ζήτηση για κρέας κουνελιών θα μειωθεί, αν δεν συμβεί κάτι. Επίσης, τα ευρωπαϊκά κονικλοτροφία δέχονται ολοένα και μεγαλύτερο ανταγωνισμό από την Κίνα. Σε αυτό προστίθεται ότι ο συγκεκριμένος κλάδος δεν λαμβάνει επιδοτήσεις στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Για όλους αυτούς τους λόγους αντιμετωπίζουμε πλέον ένα πρόβλημα επιβίωσης των ευρωπαϊκών κολυνκλοτροφίων. Και αν δεν αλλάξουμε κάτι, ο κλάδος θα εξαφανιστεί λόγω των φθηνών εισαγωγών από την Κίνα και από άλλες χώρες. Σας διαβεβαιώ ότι εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση το μερίδιο αυτό της αγοράς να το κατακτήσουν οι Κινέζοι, διότι εκεί οι μέθοδοι εκτροφής βρίσκονται πολύ πιο πίσω από αυτές που ισχύουν στην Ευρώπη. Τι μπορούμε να κάνουμε ως κοινοβούλιο λοιπόν πιστεύω ότι η μοναδική βιώσιμη ε, λύση βρίσκεται στην, ε, στον σεβασμό της ποιότητας της εκτροφής και του παραγόμενου κρέατος. Το ε, βαρόμετρο για την προστασία των ζώων που εξέδωσε την Άνοιξη η Κομισιόν έδειξε ότι πάνω από 80% των καταναλωτών ζητούν στοιχειώδεις και αξιοπρεπείς κανόνες για την εκτροφή κουνελιών. Ο καταναλωτής θέλει υψηλής ποιότητας προϊόντα τα οποία θα μπορεί να τα καταναλώνει με καθαρή τη συνείδησή του. Γι' αυτόν τον λόγο και στην έκθεσή μου επικεντρώνομαι στην ποιότητα των ε, μεθόδων εκτροφής γιατί πρόκειται για μια διαδικασία αμοιβαίου ωφέλους και για τα ζώα και για τους καταναλωτές. Από τη δική μας λοιπόν στάση εξαρτάται αν θα σεβαστούμε τις επιθυμίες των πολιτών της Ευρώπης. Ακριβώς όπως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χειρίστηκε την υπόθεση των ε, ε ορνήθων, έτσι πρέπει να ακολουθούμε, να, αυτή τη ε, διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε και στα κουνέλια. Και δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να έχει αντίρρηση σε αυτό. Ας διατηρήσουμε λοιπόν την αξιοπιστία μας και ας ε, δεχθούμε ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις κλωβοστοιχίες στα κουνέλια ενώ τις έχουμε καταργήσει ε, στα κοτόπουλα. Τότε οι επιχειρηματίες ε, εκείνου του κλάδου μας είχαν πει ότι θα τους καταστρέψουμε αν καταργήσουμε τις κλωβοστοιχίες. Ωστόσο, από το 2012 και έπειτα το αντίθετο έχει αποδεχθεί. Αν οι πολιτικοί τότε μαζί με τις επιχειρήσεις του κλάδου της ορνηθοτροφίας κατάφεραν να καταλήξουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα, τότε νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στην περίπτωση των κουνελιών. Συζητούμε πολύ αργά, θα έλεγα, για αυτούς τους στοιχειώδες κανόνες για την κονικλοτροφία. Το ΙΕΦΣΑ από το 2005 έχει ήδη διαπιστώσει ότι τα προβλήματα στην κονικλοτροφία για τα ίδια τα κουνέλια είναι πάρα πολύ υψηλά. Επιπλέον, η μαζική χρήση αντιβιωτικών στα κονικλοτροφία αποτελεί και ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, ακριβώς γιατί ήδη σήμερα χρησιμοποιούνται αντιβιωτικά ε, εξαιρετικά υψηλής δραστικότητας και που λειτουργούν συνήθως ως έσχατο, μέσος, ε, ως έσχατο μέσο. Η χρήση λοιπόν κλωβοστοιχειών αντιβιωτικών αποτελεί κακομεταχείριση των ζώων. Υπάρχουν και εναλλακτικά ε, συστήματα. Και τα προτείνω στην έκθεσή μου. Κατά τη γνώμη μου, η πρόταση που εμπεριέχεται στην έκθεσή μου εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια και την καλή διαβίωση των κουνελιών. Σε κλωβοστοιχίες κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε καμία περίπτωση. Ας μην παρασυρθούμε από δίθεν εμπειρογνώμονες ή από τους ίδιους επιχειρηματίες του κλάδου. Ο κλάδος θα έπρεπε να θεωρήσει ότι η αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας μου είναι μια ευκαιρία για τον ίδιο. Διότι στο επόμενο, το επόμενο διάστημα, με βάση και τις προτάσεις που θα λάβω, θα εμπλουτίσω την έκθεση αυτή. Η ανάπτυξη της υπαίθρου και στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να, ε, να μας οδηγήσει στο να δημιουργηθούν αξιοπρεπέστερες συνθήκες διαβίωσης και εκτροφής των κουνελιών. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό που πρέπει. Ας, κάνουμε, ας ακούσουμε τις οργανώσεις προστασίας των ζώων, ας ακούσουμε επιτέλους τους καταναλωτές που θέλουν προϊόντα που παράγονται με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και προστασίας των ζώων. Αν δεν αναλάβουμε δράση τώρα, οι Κινέζοι ανταγωνιστές θα κατακτήσουν τα μερίδια τη αγορά. Αυτά χωρίς καν να έχουμε κινηθεί εμείς προς τη σωστή κατεύθυνση. Το άρθρο 13 της συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει ότι πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά τα δικαιώματα των ζώων. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Εκ. Ποιος θέλει το λόγο. Η κυρία Γιλέρα πρώτα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Εκ για την έκθεσή του παρόλο που απέχει κάπως από τη δική μου προσέγγιση για το θέμα της κονικλοτροφίας Έχουμε μερικέ διαφορέ με τον εισηγητή, αλλά χαίρομαι για την έκθεση γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να, να μιλήσουμε για τον κλάδο αυτό. Πρόκειται για ένα κλάδο, το κλάδο τη εκτροφή κουνελιών, για τον οποίο ισχύει γενική οδηγία για, τις, ε, για την καλή μεταχείριση των ζώων. Βέβαια και η νεκροτροφία δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την οδηγία, αλλά και άλλοι κλάδοι δεν περιλαμβάνονται. Δεν είναι μόνο τα κουνέλια που δεν καλύπτονται από την οδηγία για την καλή μεταχείριση των ζώων. Έχουμε και εκτροφές άλλων ζώων που δεν καλύπτονται. Βέβαια, καλό θα ήταν να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, να περιληφθούν όλο και περισσότερα κλάδι, γιατί η συνθήκη μας ε, το υποχρεώνει είναι πολύ ενδιαφέρον ο κλάδος της κονικλοτροφίας ε, για την Ισπανία, για παράδειγμα. Ξέρω ότι ισχύουν κώδικες διοντολογίας και των πρακτικών. Εκεί υιοθετούνται όλο και περισσότερε πρακτικέ που συνάδουν με την καλή μεταχείριση των ζώων. Επίση, έχουμε μια πλατφόρμα καλή μεταχειριζών, στην οποία συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, ε, φορεί και εκπρόσωποι του κλάδου, για να ξεκινήσει μια ε, καλύτερη μεταχείριση και των κουνελιών στην κονικλοτροφία. Οπότε υπάρχουν θετικά βήματα και βελτίωση και δεν είναι τα κουνέλια το μόνο είδος που εκπίπτει του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για την ευζοία. Επίσης, η κονικλοτροφία είναι ο δεύτερος σημαντικός κλάδος εκτροφής, τουλάχιστον ως προς τον αριθμό των ζώων. Αλλά η κονικλοτροφία αντιπροσωπεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερο από το 1% της ε, τελικής ε, κτηνοτροφικής παραγωγής. Από οικονομική άποψη, αυτή είναι η σημασία του τομέα, λιγότερο από το 1%. Άλλο το θέμα της ευζοής και της καλής μεταχείρισης των ζώων. Οικονομικά πάντως είναι λιγότερο από το 1% της κτηνοτροφικής παραγωγής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, δεν είναι σημαντικός. Επίσης, ε, ε, έχετε επαφή με τον κλάδο και ξέρετε ότι και ο κλάδος βιώνει σημαντική κρίση. Και σίγουρα το θέμα της ποιότητας είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα ήθελα να αναφέρετε περισσότερο στην έκθεση την ε, ανάγκη ε, διεξαγωγής έρευνας, γιατί μιλάτε για το, τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, αλλά η θνησιμότητα αυτή είναι εγγενής ε, με το είδο αυτό, που δεν είναι και πολύ παραγωγικό και πολύ αποδοτικό. Γι' αυτό και η μεγάλη βιομηχανία δεν ενδιαφέρεται για την έρευνα στα κουνέλια. Βελτίωση της φυλής, ε, της ράτσας. Ε, ακριβώς λόγω της μεγάλης θυσιμότητας, η κονικλοτροφία δεν ενδιαφέρει τη μεγάλη ε, βιομηχανία. Πρόκειται για ένα μικρό ε, είδος, γι' αυτό και δεν υπάρχουν ειδικά αντιβιωτικά για τα κουνέλια. Όλες αυτές τις δυσκολίες αντιμετωπίζει ο εκτροφέας κουνελιών. Και με όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Και σίγουρα η ποιότητα είναι το Ειδοποιώ διαφορά ή πρέπει να είναι μεταξύ της ε, κοινοτική παραγωγής και των της υπόλοιπης παραγωγής. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα, πολύ περισσότερη έρευνα και στο θέμα αυτό και περισσότερε επενδύσει στην καινοτομία στον κλάδο της κονικλοτροφία. Βέβαια δεν έχει τόσο δυναμικό η εκτροφή κουνελιών όσο οι άλλοι ε, τομείς αλλά είναι κρίμα να μην έχουμε έρευνα για τα κουνέλια, να μην έχουμε ειδικά αντιβιωτικά για τα κουνέλια. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη έρευνα παρά τη μικρή οικονομική αξία αυτού του κλάδου. Εγώ θα ήθελα στην έκθεση να εξάρουμε ε, την ποιότητα του έργου του κονικλοτροφέα, γιατί μας ενδιαφέρει η καλή μεταχείριση των κουνελιών, αλλά θα πρέπει να αμελούμε και την ανάγκη της ευημερίας του εκτροφέα. Γιατί όπω και άλλοι γεωργικοί κλάδοι και η μας μαστίζεται από την κρίση. Γι' αυτό θα πρέπει να προτείνουμε κάποια μέτρα για να την αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν η έκθεσή μα να είναι χρήσιμη. Να ε, επιβραβεύσουμε τους κώδικες ε, βέλτισης πρακτικής και να επενδύσουμε στην έρευνα για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του κλάδου. Σας ευχαριστώ. Έχουμε μακροσκελή κατάλογο μιλητών, γι' αυτό θα αναγκαστώ να σας περιορίσω στο χρόνο. 1,5 λεπτό παρακαλώ καθένας, γιατί έχουμε πολλούς ομιλητές, πολλούς συναδέλφους που ενδιαφέρονται να λάβουν το λόγο. Λυπούμε που πρέπει να σας περιορίσω στο 1,5 λεπτό, αλλά τι να κάνουμε. Ο κύριος Λαζό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εικονοκλωτροφία, όπως ξέρετε, εκπροσωπεί 8.000 θέσεις εργασίας στην ε, Γαλλία και περίπου 1500 μονάδες. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας λοιπόν. Όπως λέμε και από άλλους ε, τομείς, ε, οι καταναλωτές δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στο πώς ε, τα ζώα θανατώνονται και φτάνουν στο πιάτο τους τα προϊόντα. Είναι πολλοί οι φορείς της κονικλοτοφίας που προτείνουν την κατάλληλη σύντηση με τα κατάλληλα προϊόντα χωρίς ε, γενετικώς τροποποιημένα ή αντιβιωτικά. Και οι καταναλωτές κρέατος που πολλές φορές ε, την κάνουν ε, μιας σκοπτικής παρουσίασης δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό. Παρόλα αυτά Βρίσκω πραγματικά ανόητες τις περισσότερες προτάσεις σας, ε, κύριε εισηγητή, ε, διότι δεν εμποδίζεται καθόλου τους εκτροφείς να συνεχίσουν την παραγωγή στις κλοβούς όπως ε, και προηγουμένως με τις ίδιες προποθέσεις και το πρόβλημα δεν είναι απλώς οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων αλλά και η καλή διαβίωση των ίδιων ακτινοτρόφων. Για τις ανάγκες λοιπόν ε, ε, σύντησης των μικρών, μικρόσωμων αυτών ζώων αλλά και προς όφελος των λίγων αυτών παραγωγών και των καταναλωτών δεν θέλουμε να υπάρχει περιοριστικός κανονισμός εδώ. Ο σκοπός είναι να καλλιεργηθούν οι καλές πρακτικές εκτροφής παρά να γίνουν υποχρεωτικές. Και επίσης πρέπει να δούμε και το κατά πόσον ε, μπορούμε να στηρίζουμε την εκτατική βιομηχανική εκτροφή και τις ε, τάσεις κερδοσκοπίας ακόμα και στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά πρώτον. Ευχαριστούμε. Κύριε Σπόλτσακ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. δυστυχώς δεν ε, κατάφερα να είμαι ε, παρόν από την αρχή της συζήτησης γιατί είχα ένα άλλο θέμα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δυστυχώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι εδώ και χρόνια αγνοεί και παραμελεί το θέμα των κουνελιών και θα πρέπει να ζητήσω μια λύση που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των πλευρών. Και ως και όδης του ΕΛΚ για το θέμα αυτό πιστεύω ότι εκτός από καλές συνθήκες στέγας και διαβίωσης ε, για τα κουνέλια εκτροφής θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν και οι καταναλωτές και τα συμφέροντα των καταναλωτών που ε, θέλουν ποιοτικό κρέας κουνελιού και κουνέλια που εκτρέφονται σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Είμαι κατά της δεσμευτικής κοινοτική ε, κοινοτικής νομοθεσίας όμως στο θέμα αυτό, γιατί για να νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχει νομική βάση στη συνθήκη που να τη δίνει τέτοιο δικαίωμα. Και αν προκειμένου δεν έχουμε νομική βάση που να εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθετικέ διατάξεις ε, για το θέμα αυτό. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δικαιούται να ε, νομοθετεί για την ευζοία ή την καλή μεταχείριση των ζώων εκτροφής, με βάση τουλάχιστον τη συνθήκη. Ο κύριος ΕΚ αναφέρθηκε στο άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μόνο όμως που λέει το άρθρο 13 είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα λάβουν υπόψη την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτό όμως είναι ένα γενικό σχόλιο ε, για τις συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα εκτροφής. και δεν αποτελεί νομική βάση για την ε, θέσπιση νομοθεσίας. Αν λοιπόν θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα διέπεται από κράτος δικαίου, θα πρέπει να αποφύγουμε ε, νομοθετικές διατάξεις για τέτοια θέματα. Επίσης, ε, μην ξεχνάτε ότι τα κουνέλια τα εκτρέφουμε για το κρέας και τη γούνα τους. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει οι κονικλοτρόφοι να επιβαρυνθούν από δυσανάλογες ε, νομοθετικές ε, διατάξεις που θα τους εξωθήσουν στην εγκατάλειψη της δραστηριότητάς τους. Δεν νομίζω ότι κανένας από εμά θα ήθελε να περιτυλίξει με τις γραφειοκρατικές διατάξεις, να εκλοβήσει τόσο γραφειοκρατικές διατάξεις στους κρονικροτρόφους, ώστε να τους αναγκάσει να εισαγάγουν κρέας κουνελιού από τρίτες χώρες που δεν έχουν τόσο υψηλές προδιαγραφές. Εκτιμώ τις καλές προθέσεις του εισηγητού του κυρίου Εκ, αλλά νομίζω ότι χρησιμοποιεί εσφαλμένες ε, δηλώσει και ασφαλμένους ε, ισχυρισμούς στο έγγραφό του. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, πρέπει να έχουμε πρώτα συζήτηση με εμπειρογνώμονες ε, ε, και να στηριχθούμε σε επιστημονικά πορίσματα και μακροχρόνιες μελέτες και έρευνες, όχι σε αισθηκτόδει αντιδράσεις και συναισθηματικές. Γι' αυτό θα καταθέσω τροπολογίες για την έκθεση. Αντιλαμβάνομαι ότι είστε ο σκιώδης ηγετής, ε, οπότε εκφέρετε και την άψη της ομάδας σας, αλλά ο χρόνος πρέπει να τηρείται για όλους. Ευχαριστώ κύριο Χόισλινγκ. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Εκ. για την ανάγκη θέσπισης κανόνων στον τομέα αυτών. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την επιχειρηματολογία του ΕΛΚ που λέει ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Ο κύριος ΕΚ επισήμανε ότι και στα Κοτόπουλα είχαμε κάνει μια αντίστοιχη ε, συζήτηση και ακριβώς επειδή θέλουμε να προωθήσουμε και να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε μας ενδιαφέρει. Ας αφήσουμε χώρες όπου ε, ισχύουν ακόμα χειρότερες προδιαγραφές από ό,τι στην Ευρώπη να έρθουν να κατακτήσουν την αγορά στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι πρέπει να θέσουμε πολύ αυστηρές προδιαγραφές και για τους ε, κτηνοτρόφους στην Ευρώπη αλλά και για τις εισαγωγές. Αν δείτε ποιες συνθήκες επικρατούν στα κονικροτροφία. Ε, δεν χρειαζόμαστε και τίποτα φοβέρες επιστημονικές μελέτες. Το κάθε κουνέλι έχει χώρο όσο περίπου μια κόλλα χαρτί α4 στα κονικλοτροφία της Ευρώπης. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχόμαστε έτσι απλά. Επίσης, μελέτες έχουν αποδείξει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση αντιβιωτικών, υπάρχουν μη καθορισμένες και πολύ μεγάλες διάρκειες μεταφοράς για τα κουνέλια και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ασχοληθούμε με αυτόν τον τομέα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε θεσπίσει νομοθεσία για όλους τους άλλους κλάδους και να αφήνουμε αυτόν απ' έξω. Και αυτό το κάνουμε και για την προστασία των καταναλωτών και για την προστασία των ζώων. Κάποιες χώρες άλλωστε έχουν ήδη θεσπίσει εθνική νομοθεσία. Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία. Πρέπει επιτέλους να κάνουμε βήματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να εναρμονιστεί ε, να εναρμονιστούν οι συνθήκες εκτροφής για τα κουνέλια στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο σας καλώ και εγώ να συνεχίσουμε το έργο μας όσον αφορά την προστασία των ζώων αλλά και των καταναλωτών και να καταλήξουμε επιτέλους στους ευρωπαϊκούς κανόνες σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα και ο κύριος Χόισλινγκ ήταν σκιώδης συγητής. Ο κύριος Άγνιο τώρα. Κύριε, ο κύριος Εκ είπε ότι τα κοτόπουλα δεν βρίσκονται στα, στους των εκτουθείων. Είστε βέβαιος διότι νομίζω ότι όταν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ρώτησε τι κυβερνήσει και τα κράτη στην Ανατολική Ευρώπη αν έχουν ακόμα κλοβούς, είπαν όχι. Δεν είμαι βέβαιος. Έχουμε αλλάξει τον ορισμό. Και οι κλωβοστοιχίες έχουν ε, αλλάξει η παραγωγή συνεχίζουν να πουλάνε στην Ανατολική Ευρώπη, οπότε κατά πάσα πιθανότητα απλώ συνεχίζουν να υπάρχουν. Και για τα κουνέλια. Εδώ, ε, για το άρθρο 13 τη συνθήκη, είπε κάποιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικαίωμα να μοθετήσει σε αυτό το τομέα. Και παρόλα αυτά υπάρχει μια διάθεση να συνεχίσουμε. Μετά ποιοι θα ακολουθήσουν, τι ποια ζώα θα ακολουθήσουν, στροφοκάμελοι και τα λάμα. Υπάρχει κάτι για το οποίο δεν έχει νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί σε κάθε περίπτωση στη χώρα μου έχουμε νομοθεσία για την εκτροφή των κουνελιών και δεν θέλουμε να υπάρξει επικάλυψη με ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, Πρόεδρε, ελπίζω ότι σα γλίτωσα κάπω ο χρόνο. Να με ευχαριστείτε. Σα ευχαριστούμε θερμά. Διπλά. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Χάζεκάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Εκ για την έκθεσή του, για την εκτροφή των κουνελιών. Είναι ένας τομέας ο οποίος αξίζει όλη μας την προσοχή. Πρόεδρε, ήθελα να θίξω δύο σημεία, τα οποία θεωρώ ότι είναι ζήτημα παρανόησης. Ε, το πρώτο, πρόκειται για ένα τομέα αρκετά περιορισμένο. Δεν έχει ανάγκη να νομοθετήσουμε γι' αυτόν και θα δυσκεράνουμε τη ζωή των εκτροφέων. Αυτό λέει και ο κύριος Τίμερμανς ε, γενικώ για πολλά άλλα θέματα πέραν αυτού. Και η δεύτερη, το δεύτερο σημείο παρανόησης που θέλω να θίξω είναι ότι είναι ένα τομέα στον οποίο δεν αξίζει να επικεντρωθούμε γιατί υπάρχουν άλλοι πολύ σημαντικότεροι που θα άξιζαν περισσότερο την προσοχή μας. Θα ξεκινήσω με την τελευταία παρατήρηση. Η εκτροφή κουνελιών είναι ένας κλάδος που δεν ε, έχει να κάνει δεν είναι κάτι που έχουν αναλάβει πιο εθεροβάμονες από τους κοινοτρόφους μας. Εδώ πρόκειται για κάτι το υπαρκτό. Τα ζώα, ε, τουλάχιστον υπό το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας, είναι πλάσματα ευάλωτα. Πρέπει να τα προστατεύσουμε. Ε, θα πρέπει λοιπόν οι κανόνες να ισχύουν με τρόπο παρόμοιο για όλα τα ζώα, είτε είναι ζώα συντροφιάς και ασχέτως της σημασίας του κλάδου που εκπροσωπούν από την πλευρά των κτηνοτροφικών εισοδημάτων. Οι κανόνε, λέει κάποιο, δεν είναι αναγκαίοι και θα πρέπει να αυτορυθμιστεί ο όλο τομέα και να προστατεύουν οι ίδιοι οι εκτροφεί στα ζώα του. Δεν είναι έτσι. Πρόεδρε, στην εκτροφή κουνελιών έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε να επαφιόμαστε στην καλή διάθεση των εκτροφέων Εάν μόνο πρόκειται για ζώα, δηλαδή με ψυχαγωγικούς σκοπούς, κοινωνικούς, ε, να τα προστατεύουμε, ιδάλλως όχι. Ακόμα χρησιμοποιούνται κλωβοί. Τα ζώα δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να παίξουν και ε, γι' αυτό χαιρετίζουμε την έκθεση αυτή. Και ελπίζω οι συνάδελφοι να σκεφτούν πολύ σοβαρά το κατά πόσο να ε, δει να ασχολείται η υποτροπή μας με ένα τέτοιο θέμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να μιμηθείτε το παράδειγμα του κυρίου Άγγινιου ό,τι αφορά το χρονογόρευση. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα αυτό. Και αντίθετα με αυτό που ακούσαμε στην αρχή, το θέμα της οικονομίας και της οικονομικής διάστασης της κονικλοτροφίας είναι σημαντικό για αρκετές χώρες, κυρίως ε, της Νότιας Ευρώπης. Και είναι σημαντικό να συζητούμε αυτά τα θέματα. Τώρα, για την έκθεση καθευτή. Παρά είναι επικεντρωμένη έκθεση στο θέμα σε δύο πτυχές της κονικολοτροφίας. Και μάλιστα είναι μερικές φορές στο περίπου σε ό,τι φορά κάποιους ισχυρισμού. Μάλιστα μερικές φορές περιέχει και ανακρίβειες, ιδιαίτερα στο μέγεθος των κλοβών. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μία έκθεση πυρογνωμόνων της ΕΦΣΑ του 2005 που έδειχναν ότι οι διαστάσεις των κλοβών ήταν σημαντικές και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την άνεση των ζώων και την υγιεινή των ζώων. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμα τα σχόλια που έχετε για τις συγκεκριμένες διαστάσεις και πόσο η, τα χαρακτηριστικά των κλοβών μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοια ταλαιπωρία των ζώων. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κορυκλοτροφίας. Και ε, σωστά αυτό που μας είπε η κυρία Αγγιλέρα. Επίσης, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους κορυκλοτρόφους για να εξελιχθούν και να εφαρμόσουν καλύτερα συστήματα όπως αυτό το περιφράγματος γιατί κάτι τέτοιο εξυπηρετεί και την οικονομική λογική αλλά και τη λογική της καλής μεταχείρισης των ζώων και άρα και των ίδιων των εκτροφέων. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξελιχθούμε σε πολύ πιο πρόσφατα πορίσματα και επιστημονικές μελέτες. Ευχαριστώ. Κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, και κυρίως ο κύριος Ανδρία πριν από λίγο, η παραγωγή κρέατος κουνελιού είναι σημαντική για αρκετές χώρες, ιδιαίτερα της Νότιας Ευρώπης και ανταποκρίνεται σε μια γαστρονομική παράδοση πολλών περιφερειών. Και διάβασα με μεγάλη προσοχή την έκθεση του κυρίου Εκ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι η έκθεση αυτή εκπονήθηκε μετά από διαβουλεύσεις ε, με εκπροσώπους από ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Νομίζω ότι ε, επικεντρώνεται σε μια πολύ μονομερή προσέγγιση, γιατί η εικονικλοτροφία είναι κάτι δύσκολο, γιατί το κουνέλι είναι πολύ ιδιαίτερο ζώο από βακτηρολογική κυρίως άποψη. Οπότε πρόκειται για ένα α, ζώο που έχει κοινωνική ζωή, αλλά είναι και αρκετά επιθετικό. Ε, γιατί έχω και εγώ προσωπική εμπειρία από κονικλοτροφή και ξέρω πόσο οι καυγάδες μεταξύ των ζώων ε, μπορούν να προκαλέσουν ζημιές ε, λόγω της επιθετικότητας. Οπότε θα πρέπει να επανισορροπήσουμε την έκθεση γιατί παρά είναι μονόπλευρη και ίσω μεροληπτική και να λάβει με υπόψη με την έκθεση ένα ευρύτερο φάσμα απόψεων και κυρίω να λάβουμε υπόψη τα τελευταία επιστημονικά πορίσματα και τι πιο πρόσφατε επιστημονικέ μελέτε. Νομίζω ότι χάρη σε τέτοιε πιο επικαιροποιημένε μελέτε θα καταστήσουμε πιο ρεαλιστική την έκθεση. Σα ευχαριστώ κύριο Ντενανό. Πρόεδρε, η έκθεση σίγουρα αξίζει να επιβάλλουμε πολλακίες για να την εξορροπήσουμε σωστά. Όμως, Νομίζω ότι αντιθέτως με αυτό που λένε κάποιοι εδώ, είναι προς τιμή του Κοινοβουλίου να ασχοληθεί με ένα τέτοιο θέμα, την εκτροφή των κουνελιών. Ε, και βεβαίω είναι τιμή και για την Επιτροπή μα. Είναι ένα σοβαρό το θέμα, είναι θέμα δημόσια υγεία, είναι θέμα ποιότητα του κρέατο που παράγουμε, με όλου του προβληματισμού ε, περί αντιβιωτικών που υποκρύπτει η εκτροφή κουνελιών, ε, αντιβιωτικά που εν γέννη μα απασχολούν και πολύ συχνά έχουν βλαβερέ συνέπειε. Δεύτερο σημείο, που υπονοείται εδώ είναι βεβαίω η καλή διαβίωση των ζώων και δεν ξέρω αν έχουμε επιλύσει το θέμα των ε, κοτόπουλων που πρόκειται να σπαγιαστούν να καταναλωθούν, αλλά Πραγματικά μετά την επίσκεψή μου στο σφαγείο έχω μεγαλύτερο πρόβλημα να φάω κρέα από κοτόπουλο. Σκεφτείτε τα λοιπόν σοβαρά αυτά, γιατί έχουν πραγματικά να κάνουν με την καλύτερη διαβίωση των ζώων. Και τρίτο θέμα που πολλέ φορέ τέθηκε, είναι ένα τομέα που έχει οικονομικά κέρδη. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από την εκτροφή κουνελιών. Οπότε είναι σημαντικό οι εκτροφεί να μπορούν να ζουν από αυτό που παράγουν και να έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ευχαριστούμε κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο ΕΚ για την έκθεσή του, για το σχέδιο έκθεσης. Και εγώ πιστεύω ότι η έκθεση αυτή αξίζει να συζητηθεί και πρέπει κατά κάποιο τρόπο να πάρουμε θέση, να παρέμβουμε. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν μόλι από άλλου συναδέλφου. Πρέπει να προσέξουμε και να δώσουμε σημασία στην καλή διαβίωση των ζώων, να βελτιώσουμε την υγεία του. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να μιλήσουμε και για το συμφέρον, για τα ωφέλη δηλαδή, όσων ασχολούμαι με αυτόν τον οικονομικό τομέα. Είναι λοιπόν νομίζω ανάγκη να νομοθετήσουμε στο θέμα αυτό. Οι καταναλωτέ δίνουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή και κοιτάζουν να ψάξουν τις συνθήκες εκτροφής των ζώων. Τις ελέγχουν. Ένα σημείο που δεν φύγεται στην έκθεση και νομίζω καλό να εντοπιστεί είναι αυτό της ε, επισήμανσης. Πρέπει να δούμε μήπως πρέπει να υπάρχει και ένδειξη προέλευσης του κρέατος, όχι μόνο ο τόπος σφαγής. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα αποφύγουμε η αγορά μας να κατακλειστεί και από κρέατα έξω ευρωπαϊκά. Σε ό,τι αφορά την εκτροφή και τις συνθήκες που θα πρέπει να γίνουν πρότυπο, ε, θα συμφωνήσω με τον κύριο Αντριέ. Πρέπει να διευκολύνουμε τις νέες μορφές εκτροφής που μπορεί αναντήρητα να περιορίζουν τη χρήση αντιβιωτικών που βλάπτουν τόσο πολύ ακόμη και την ανθρώπινη υγεία. Ευχαριστώ. Κυρία Μίλλερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ τον σκιώδη εισηγητή μας, τον κύριο Ρόντε. Είναι φυσικά πολύ σημαντικό να θεσπιστούν στοιχειώδες κανόνες για να εξασφαλιστούν ίση όρια ανταγωνισμού για τους παραγωγείς, ακριβώς γιατί οι, ανταγων... οι επιχειρήσεις δέχονται ανταγωνισμό από την Κίνα. Επίσης θα πρέπει να καταργηθούν οποιασδήποτε μέθοδοι κακομεταχείρισης των ζώων. Έχουν ήδη ε, ληφθεί τέτοια βήματα σε διάφορα κράτη, ε, μέλη και φυσικά ε, ο σκιώδης μας συμφωνεί όσον αφορά την ανάγκη προστασίας των ζώων. Η Κομισιόν θα μπορούσε με νομοθετικές της προτάσεις να κλείσει αυτό το νομοθετικό κενό. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε το πώς θα χειριστούμε αυτό το θέμα και εμείς ως ΑΛΔΕ θα συνεργαστούμε στενά με τον εισηγητή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα σταλεί το σωστό μήνυμα τόσο προς την Κομισιόν όσο και προς τον κλάδο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η ευημερία των ζώων αλλά και ε, τα οικονομικά συμφέροντα του κλάδου και βεβαίως θα μπορούσαν ε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο σε ορισμένα κράτη-μέλη να λειτουργήσουν ως οδικός χάρτης για τους κανόνες που θα μπορούσαν να θεσπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διπλά ευχαριστώ που και σύντομοι. Κυρία Νόιχλ. Ε, Εγώ θέλω να υποστηρίξω την, ε, το σχέδιο έκθεσης του κυρίου ΕΚ. Το κάνω, μόνο, το κάνω και εκ μέρους της κυρίας Κάραν Κάτεμπαφερ. Νομίζω ότι η έκθεση δείχνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί στην Ευρώπη έχουμε σοβαρότατα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Πρέπει να θεσπιστούν στοιχειώδεις δεσμευτικοί κανόνες για την κονικλοτροφία. Είναι μια απέτηση που έχουν οι ψηφοφόροι μας και οι καταναλωτές στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο ε, άλλοι βεβαίως μιλούν για γαστρονομικές παραδόσεις, άλλοι μιλούν για κρέατα, για δέρματα, για γούνες. Εγώ όμως θα κάνω λόγο για ζώα. Εγώ τρώω κρέας, δεν έχω πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να θεσπιστούν στοιχειώδεις τουλάχιστον κανόνες για την εκτροφή των κουνελιών. Αναφέρθηκε το ζήτημα των, ε, της ορνηθοτροφίας τότε οι επιχειρήσεις του κλάδου έλεγαν ότι θα μας καταστρέψετε με αυτούς τους κανόνες. Δεν έγινε όμως ποτέ κάτι τέτοιο. Έπειτα από μια μακρά μεταβατική περίοδο ο κλάδος βρίσκεται σε διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης. Κατά τη γνώμη μου ε, ε, ε, στην Αυστρία, τη χώρα από την οποία κατάγομαι, υπάρχουν ήδη ελάχιστοι ε, κανόνες και αυτοί θα πρέπει να διευρυνθούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, σε εμάς ε, απαγορεύονται τα σειρματοπλέγματα, οι κλωβοστοιχίες, υπάρχει επαρκής χώρος για τα ζώα. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται και να στεγάζονται τα ζώα το ένα πάνω από το άλλο. Ε, πρέπει να έχουν επαρκή πρόσβαση σε νερό και τροφή και φυσικά θα πρέπει να ανισθητοποιούνται πριν από, την, ε, πριν από τη θανάτωσή τους. Αυτές οι προδιαγραφές πρέπει να επεκταθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και μια ένωση αξιών, που βέβαια δεν αφορούν μόνο την ευημερία των ζώων, αλλά ένα ευρύτατο φάσμα ε, ανθρώπινης ο κλάδος πρέπει να κατανοήσει ότι αυτή η θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών είναι μια ευκαιρία για τον κλάδο. Γιατί θα ισχύουν οι ίδιες ε, προδιαγραφές και για τις εισαγωγές. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αποκρούσουμε και τις φθηνές εισαγωγές από την Κίνα. Ε, η σκιώδη συγγήτρια την οποία σήμερα εκπροσωπώ ε, θα υποβάλει πρωτοτροπολογίες για την καθαριότητα, για την επιτήρηση και για την αναισθητοποίηση και για μια σειρά άλλα θέματα. Επίσης θα ήθελα προσωπικά να ε, κάνω μια παρατήρηση. Δεν είναι της σκιώδης συγγήτριας. Το γεγονός ότι οι διάφοροι οικονομικοί κλάδοι αισθάνονται ότι δέχονται πιέσεις είναι γεγονός. Γι' αυτό και βλέπουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα των λόμπι και των ε, επιστολών που μας αποστέλλονται. Εμείς όμως πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν θέλουμε να τους καταστρέψουμε ούτε να καταργήσουμε την κονικλότροφία στην Ευρώπη. Θέλουμε αντιθέτως να συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά θα πρέπει στην, στο μέλλον η επιχειρηματική τους δραστηριότητα να χαρακτηρίζεται από την προστασία της αξιοπρέπειας των ζώων για να μπορούν και οι καταναλωτές με καθαρή τη συνείδησή τους να καταναλώνουν τα προϊόντα τους. And, uh, first... Ο Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα τον κύριο Στέφανάκη για την έκθεσή του. Μερικές φορές ε, ε, ε, εδώ στο Κοινοβούλιο είναι σαν να με ρωτάνε μια μέρα που βρέχει που καταφέρα και βρέχτηκα. Τι θέλετε, επιστημονικές μελέτες, όταν ε, κουνέλια σε τα εκτρέφουμε σε τέτοιες συνθήκες. Ε, σταθείτε με μία εβδομάδα σε τόσο στενό χώρο και θα δείτε αν θα ζητάτε μετά μελέτες για να αποδεικνύετε πόσο βασανιστικό είναι να εκτρέφονται κουνέλια σε τόσο ε, στενός ε, κλωβοστοιχίες. Βέβαια, κάποιο από την Ιρλανδία δεν πρόκειται να πει σε κάποιον από τη Γαλλία τι πρέπει να κάνει. Πάντω, αν εγώ ζούσα στην Γαλλία ή αν ζούσα στην Ισπανία, δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω με τίποτα από όσα αναφέρονται στην έκθεση. Γιατί ο κύριος Δενανό είπε κάτι πολύ εύστοχο, ότι όταν ε, επισκέφθηκε κλωβοστοιχίες ε, με κοτόπουλα δεν είχε πια διάθεση να καταναλώσει κρέας ε, κοτόπουλου. Αυτό θα πρέπει να ενδιαφέρει την βιομηχανία. Και αν θέλει να καταπολεμήσει τις αγωγές από την Κίνα θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και διαφοροποιείται με την καλύτερη ποιότητα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Δενανό. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Εκ για την έκθεσή του και ίσως δεν είναι αρκετά ευρεία η έκθεση και ίσως είναι κάπως μονόπλευρη. Αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε ίσως. Δεν ξέρω όμως πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε μια τέτοια έκθεση. Καλύτερα να αφήσουμε αυτά τα θέματα στις εθνικές αρχές παρά να τα ρυθμίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μερικοί αναφέρθηκαν σε κλωβοστοιχίες και συνέκριναν ε, την κατάσταση με τα κοτόπουλα. Τα, οι κλωβοστοιχίες όμως ε, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυγών, όχι για την παραγωγή κρέατος κοτόπουλου. Θα πρέπει λοιπόν να εμείνουμε στα πραγματικά περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόσφατα είχαμε μία απόφαση μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Και παρόλο που εμεί δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη την απόφαση για τα σκλαβοστοιχεία. Και όταν είχαμε υποβάλει την απόφαση για τις εμπλουτισμένες κλωβοστοιχείες, τα, τα σούπερ μάρκετ, αποφάσισαν από το 2025 να μην πουλούν αυγά που προέρχονται από κλωβοστοιχείες, όσο εμπλουτισμένες και αν είναι. Δεν περίμενα λοιπόν το σούπερ μάρκετ ε, την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει απαγόρευση τέτοιων τρόπων εκτροφής για παραγωγή αυγών. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε πολύ ε, ταραγμένα νερά και σκάβουμε το λάκκο μας με την υπερβολική νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κινδυνεύουμε θεσπίζοντας υπερβολικές νομοθετικές διατάξεις. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, στον κύριο Σιμόνο, από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΜΚΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός, διότι πολλά ήδη υπόθηκαν και είναι και ορθά. Δεν θα τα επαναλάβω. Απλώς να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή και παρακολουθεί για να δει ποιο θα είναι το τελικό περιεχόμενο της ε, έκθεσης. Μα ενδιαφέρει, όπω είπα, και η συζήτηση όμω για το περιεχόμενο προηγουμένω, Ένα πράγμα που ανέκαθεν λέγαμε είναι ότι δύο αρχέ, που συμπεριλαμβάνει και η συνθήκη είναι οι εξή. Οι αρχέ τι οποίε πρέπει να βασιζόμαστε. Επικουρικότητα και αναλογικότητα. Για τι δύο αυτέ αρχέ πρέπει να μελετήσουμε σαφώς το τι θα θελήσουμε να προκρίνουμε με μια τέτοια έκθεση. Κάτι άλλο που πρέπει να πω είναι ότι ως προς την καλή διαβίωση των ζώων σήμερα, η Επιτροπή ως τώρα έχει μια οριζόντια προσέγγιση περισσότερο που να βασίζεται περισσότερο στο διάλογο, τη συζήτηση και την ανταλλαγή, την πληροφοριών και όχι στην νομοθεσία. Δηλαδή η προσέγγιση για την δημιουργία πλατφορμών λόγου χάρη που σήμερα λείπει και το έχει εντοπίσει και ο Επιτροπός μας είναι μια καλή επιλογή. Έπειτα, μετά από την πολιτική συμφωνία και τον κανονισμό για του επίσημου ελέγχου που ολοκληρώθηκε αυτό το καλοκαίρι, υπάρχει και ένα άλλο σύστημα πέραν αυτού του κανονισμού που είναι τόσο περίπλοκο, αλλά με δύο συγκεκριμένα άρθρα ω προ την καλή διαβίωση των ζώων. Αυτά θα είναι σημείο αναφορά για την καλή διαβίωση των ζώων στην Ευρώπη. Βεβαίω θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα ένα χρόνο μέχρι να εγκριθεί επισήμω ο κανονισμό. Τα δύο αυτά μέτρα, δηλαδή οι πλατφόρμε λόγου χάρη και η δημιουργία ενό κέντρου ή πολλών κέντρων αναφορά για την καλή διαβίωση των ζώων, είναι μέτρα που μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάγκη να καλύψουμε και τις ανάγκες ειδών που δεν είναι τόσο σημαντικά από οικονομικής άποψης ίσως, αλλά των οποίων μπορούμε να βελτιώσουμε την περαιτέρω τις συνθήκες διαβίωσης. Ευχαριστούμε. Κύριε Εκ, ε, ο εισηγητής μας τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω σε ορισμένα από τα επιχειρήματα που ακούστηκαν. Πολύ σύντομο. για την κυρία Γκουγέ. Εδώ και 20 χρόνια υπάρχουν έρευνες για την κονικλοτροφία. Εγώ, μάλιστα, έχω μιλήσει με τη γερμανική κυβέρνηση ήδη από το 1997. Τότε μου είχαν πει ότι ξεκινούμε τις έρευνες. Μετά από πέντε χρόνια μου είπαν το ίδιο. Και άλλα πέντε χρόνια μετά ακόμα γίνονταν έρευνε. Και σήμερα αν ρωτήσετε πάλι έρευνε γίνονται. Ειλικρινά απορώ, τι, τι ερευνούν τόσα χρόνια. Ένα ζώο που έχει την φυσική διάθεση να κινείται στο φυσικό του περιβάλλον. Δεν χρειάζεται έρευνες για να πούμε ότι δεν μπορούμε να το έχουμε σε κλουβιά του μεγέθους μιας κόλλας χαρτιού. Εγώ δεν δαιμονοποιώ τον κλάδο. Αντιθέτως, όπως είπα και εισηγητικά, θεωρώ ότι θα πρέπει να θεωρήσουν ότι αυτή η έκθεση είναι μια ευκαιρία για να μπορέσει ο κλάδος να επιβιώσει στον διεθνή ανταγωνισμό. Δεν θέλω να παραδώσουμε το μερίδιο αυτό της αγοράς στους Κινέζους. Αντιθέτως, πρέπει με υψηλές προδιαγραφές προστασίας των ζώων και προστασίας των καταναλωτών να θέσουμε εκείνους τους κανόνες προκειμένου ο ίδιος ο κλάδος να μπορέσει να, επιβιώσει. Λαζό, ο κλάδος φταίει για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Διότι εδώ και δεκαετίες δεν έκανε απολύτως τίποτα. Το σφάλμα είναι, δική, είναι δικό τους. Υπήρξαν επιχειρήσεις βιολογικής γεωργίας που υπέδειξαν στον κλάδο πώς θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη εκτροφή, αλλά ο κλάδος τους αγνόησε. Ο κύριος Πόλτσακ δυστυχώς δεν παρακολούθησε την εισαγωγική μου ομιλία, γιατί θα είχε διαπιστώσει ότι με ενδιαφέρουν πολύ και τα συμφέροντα του κλάδου. Αλλά το να λέει ότι δεν υπάρχει ανάγκη θέσπισης κανόνων, μα γιατί να μην υπάρχει τέτοια ανάγκη, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει. Το κάναμε στα, στα, το κάναμε στα κοτόπουλα, το κάναμε στα μοσχάρια. Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι για τα κουνέλια δεν χρειάζονται κανόνες. Μα έτσι στην ουσία επιτίθεται στους συναδέλφους του που ε, για χρόνια ολόκληρα αγωνίζονταν να θεσπιστούν κανόνες για τα άλλα ζώα. Εγώ θα έλεγα ότι εκείνος μεροληπτεί, όχι εγώ. Για τον κύριο Νταντών. Είπε ότι τα ζώα αυτά ε, δαγκώνουν το ένα το άλλο, επιτίθενται το ένα το άλλο. Κύριε Νταντών, αυτό συμβαίνει όταν κανείς αναγκάζει ζώα να συνεπάρχουν σε τόσο μικρό χώρο. Το ίδιο θα συνέβαινε και σε άλλα ζώα, θα συνέβαινε και σε, και ποντίκια και σε αρουραίους. Διότι πανικοβάλλονται τα κουνέλια μέσα στα κλουβιά αυτά. Γι' αυτό επιτίθενται το ένα στο άλλο. Ενώ στα συστήματα με περιφράγματα τέτοιου είδους φαινόμενα είναι πολύ πολύ λιγότερα. Θέτω λοιπόν ένα τεράστιο ερώτημα στην παρατήρησή σας να επανέλθω στην, ε, στην, στην πραγματικότητα. Εσείς θα έπρεπε να επανέλθετε στην ε, πραγματικότητα. Οι τραυματισμοί συμβαίνουν ακριβώς λόγω της έλλειψης χώρου. Μια ερώτηση προς, τον, ε, προς την Κομισιόν. Εγώ μίλησα πριν από κάποιους μήνες με τον ίδιο τον κύριο Άντριου και μου είπε εκείνος ότι είναι σημαντικό να κλείσουμε τα κενά αυτά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν είναι δυνατόν να, να υπάρχουν κανόνες για όλα τα εκτρεφόμενα ζώα και να αφήσουμε αυτό το κενό για τα κουνέλια. Μου είπε ο κ. Ανδριουκάητης ότι πρέπει να το κλείσουμε αυτό το κενό. Ε, αυτό το κενό μπορούμε να το κλείσουμε μόνο αν θεσπίσουμε κανόνες που θα ισχύουν με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Στην Αυστρία υπάρχουν κανόνες και σε κάποιες άλλες χώρες επίσης έχουν ήδη θεσπιστεί κανόνες. Μα αν δεν θεσπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κανόνες, τότε θα στρεβλωθεί ο ανταγωνισμός. Να ευχαριστήσω και για την κυρία Νόιχλ ε, για τις παρατηρήσεις που υπέβαλε και εκ μέρους της Κάντερμπαχ. και την, ευχαριστώ και την κυρία Μιούλερ που είπε ότι δεν είμαστε μόνο μια οικονομική ένωση αλλά είμαστε μια ένωση αξιών και θα πρέπει ακριβώς για αυτόν τον λόγο να αποτελέσουμε και το πρότυπο για τον κόσμο αλλά και για τους πολίτες μας. Διότι αν οι πολίτες μας διαπιστώσουν ότι εδώ οι πολιτικές ελίτ αγνοούν τις επιθυμίες των ψηφοφόρων και των πολιτών, τότε Βρισκόμαστε στο λάθος δρόμο, γιατί θα ενισχύσουμε την εικόνα ότι υπάρχει διαπλοκή και υπάρχει διαφθορά στα υψηλά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως θα πρέπει να πάρουμε και αυτό υπόψη μας, ιδίως αυτοί που λένε ότι ε, καθόμαστε και σχολιόμαστε με τα φτωχά κουνελάκια. Εν πάση περιπτώσει αυτά ε, είχα να πω εγώ από την πλευρά μου. Χαίρομαι για το έργο που έχουμε μπροστά μας με τους σκιώδεις και νομίζω ότι μπορούμε ο καθένας από την ε, σκοπιά του να βάλει ένα μικρό λιθαράκι για την προστασία των ζώων και των καταναλωτών και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να διαβούμε αυτό το, το δρόμο που έχουμε μπροστά μας και να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα για όλες τις πλευρές. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κατά νου το καλό του κλάδου, αλλά και την καλή μεταχείριση των ζώων. 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι λίγη η προθεσμία για τις τροπολογίες, η έγκριση ε, θα γίνει το Νοέμβριο, η ε, έγκριση. 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, 12 το μεσημέρι, λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες. Περνάμε τώρα στην παρουσίαση της έκθεσης ε, του Τμήματος Πολιτικών για τις αλληλεπιδράσεις της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με την κοινή γεωρική πολιτική. Όπως ξέρετε, ε, είχαμε σταδιακές εξελίξεις της κοινή γεωρικής πολιτικής. Έγιναν αρκετές μεταρρυθμίσεις. Η κοινή γεωρική πολιτική επηρεάζεται και από εξωτερικούς παράγοντες που αποκτούν όλο και περισσότερη βαρύτητα, ιδιαίτερα μετά την παγκοσμιοποίηση και την αλληλεπίδραση της παγκόσμιας αγοράς με την ευρωπαϊκή. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν την κατάσταση του Γεωργού, την κοινή γεωργική πολιτική, αλλά διαμορφώνουν και δημιουργούν και νέες προκλήσεις για την κοινή γεωργική πολιτική και αυτές θα πρέπει να λάβει υπόψη η κοινή γεωργική πολιτική στις νέες της μεταρρυθμίσεις. Ε, άλλωστε έχουμε πολλές διαπραγματεύσεις εμπορικές ε, με το Μερκοσούρ, το TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείε. και λογικό είναι και σε αυτές να λαμβάνουμε υπόψη την ιδιαίτερη θέση της Γεωργίας. και να μην χρησιμοποιηθεί η, Γεωργία ως εξυλαστήριο θύμα ή να μείνει ξεχασμένη σε τέτοιου είδου διαπραγματεύσει. Ο κύριος Σουίμπανκ ε, θα μας παρουσιάσει την ε, μελέτη αυτή από το Τμήμα Πολιτικών. Είναι καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου του Ρέντινγκ και παρακαλώ κύριε Σουίμπανκ, περιμένουμε την μελέτη σας. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, thank you, Mr. Chairman, for those words of... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα εισαγωγικά σας λόγια. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση σήμερα. Τίτλος της έκθεσης. Αρκετά ακριβής. Αλληλεπίδραση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τη κοινή γεωργική Πολιτική. Το πρώτο που θα προσθέσω να κάνω είναι να εξηγήσω τη συλλογιστική μου στην οποία βασίστηκε και η έκθεση. Μετά θα παρουσιάσω τα περιεχόμενά της. Είναι μακροσκελής η έκθεση, θα ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό. Και το βασικό ε, θέμα της παρουσιασής μου θα είναι κυρίως τα σημεία τα οποία επέλεξα και ξεχώρισα για να σας παρουσιάσω ως βασικότερα από τα πορίσματα, παρά να σας κάνω την πλήρη επισκόπηση. Και μετά θα ολοκληρώσω με τις εξωτερικές δράσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την, αγροτική, την κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2020. Ποιο είναι λοιπόν το θέμα της έκθεσης. Μου ζητήθηκε να διερευνήσω πώς οι εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επηρεάσει την κοινή αγροτική πολιτική. Διαφέρει αυτό το αντικείμενο από αυτό άλλων προηγούμενων εκθέσεων, από το κατά πόσον συνάδει με τις εξωτερικές δράσεις ε, η, της Ευρωπαϊκής Ένωσης η, η ΚΑΠ συνήθως. Ήταν το αντικείμενο. Υπήρξαν πολλά επικριτικά σχόλια, ιδίως για την παλαιότερη ΚΑΠ και τον τρόπο που είχε επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σκοπός της έκθεσης αυτής ήταν να μελετήσει ποιες είναι οι εξωτερικές επιδράσεις στην ΚΑΠ. Το δεύτερο γενικό σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι προφανώς η ΚΑΠ του 2016 διαφέρει από την αρχική ΚΑΠ όπως είχε διοργανωθεί πριν από πολλά χρόνια. Και αν κανεί παρατηρήσει τα στάδια εξέλιξη της ΚΑΠ, πολύ συχνά θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν ε, συσχετισμοί με τις ε, εξωτερικές εξέλιξει και τι αλλαγές που επιφέρθηκαν στην ΚΑΠ. Τώρα, αν το αίτιο ήταν οι εξωτερικέ αλλαγέ, ή ήταν απλώς συμπτώσει και συγκυρίε, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρουμε αν τα πράγματα θα είχαν πάει διαφορετικά εφόσον δεν υπήρχαν αυτέ οι εξωτερικέ εξέλιξει και επιρροέ. Εάν δει λοιπόν, αν δει λοιπόν κανεί τι έγινε πριν από 30 και 40, εδώ και 30 και 40 χρόνια σχεδιασμού πολιτική, είναι πολύ δύσκολο να πούμε εάν οι αλλαγέ προκάλεσαν ε, τι μεταρρυθμίσει τη ΚΑΠ ή αντίστροφα. Επίση, οι πυλώνε 1 και 2 οι μέθοδοι στήριξη τη ΚΑΠ έχουν αλλάξει πολύ, όπω ε, και η εμπορική της πολιτική, οι εμπορικοί μηχανισμοί. Ασχολείται λοιπόν η έκθεση με φυτογειονομικά μέτρα ή την καλή των ζώων, αλλά όχι μόνο, διότι αλλιώ θα είχαμε μια πολύ περιορισμένη εικόνα τη ΚΑΠ. Όπω είπα, η έκθεση είναι μακροσκελής. Εδώ σα έχω απλώ ένα κατάλογο με του τίτλου των βασικών κεφαλαίων αν θέλετε να πάρετε μια γεύση απλώς και μετά να πάτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες της έκθεσης, το κεφάλαιο 2 αφορά τρεις βασικές εξελίξεις στην ΚΑΠ. Το 92 ε, την αλλαγή στα, στην αγορά κερασιών, μετά την κοινή αλληλευτική πολιτική και μετά την θέσπιση της πολιτικής της υπαίθρου. Το τρίτο κεφάλαιο είναι η ουσία της έκθεσης, διότι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω είναι ότι οι εξωτερικές πιέσεις με την πρώτη Γενική Συμφωνία για τις ε, τιμές και τους δασμούς ήταν ε, το πρώτο στοιχείο που έφερε και άσκησε επιρροή για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΤ τα προηγούμενα χρόνια. Οι κανόνες του ΓΚΑΤ, της Συμφωνίας ΓΚΑΤ, έχουν να κάνουν με όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια που αναπτύσσω στην ε, έκθεση αυτή. Να ξεχωρίσω τώρα κάποια βασικά πορίσματα, αντί να σας ε, εξηγήσω όλους τους τίτλους όλων των κεφαλαίων, βήμα-βήμα. Και εγώ ίδιος ευνηδιάστηκα όταν κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η ΚΑΠ έχει επηρεαστεί πολύ περισσότερο από την εξωτερική πίεση από ό,τι θα μπορούσε κανείς αρχικά να υποθέσει. Εγώ μελετώ την ΚΑΠ εδώ και πολλά χρόνια. Δούλευα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από 40 χρόνια. Δεν είναι... Ε, λες και αυτά τα γεγονότα τα πήρα χαμπάρι. Όμως, πραγματικά η πίεση είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχα συνειδητοποιήσει. Ένα βασικό θέμα που διατρέχει όλα μου τα συμπεράσματα είναι το κατά πόσο η συμφωνία ΓΚΑΤ, ε, οι διαπραγματεύσει τη Ουρουγουάης και τη Ντόχα, ε, του ΠΟΕ, έχουν επηρεάσει την ΚΑΠ. Δηλαδή, η μεταρρύθμιση του 1992 επηρεάστηκε πάρα πολύ από τις διαπραγματεύσεις της Ουρουγουάης, όπως και η αλληλευτική πολιτική ε, η έννοια της αποσύνδεσης. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το κύριο της Δόχας. Άλλωστε, ήδη πολύ έχετε αναφέρει πόσο περισσότερη συνδεδεμένη βοήθεια θα θέλατε για το μέλλον. Είναι ένα από τα βασικά μα θέματα αυτά. Ή επίση οι διαδικασίε επίλυση διαφορών. Ε, Α θυμηθεί κανεί τη μεταρρύθμιση του τομέα τη ζάχαρη το 2005 και 2006 είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου η εξωτερική πίεση πραγματικά έφερε τη μεταρρύθμιση εσωτερικώς. Υπάρχουν όμως και άλλες διατάξεις της συμφωνίας GATT που επηρεάζουν την εμπορική μας θέση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, όπως το άρθρο 24 που διέπει τις συμφωνίες του ΕΟΧ, μάλλον του χώρου ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών. Εάν δούμε τώρα το πώς έχει επηρεάσει η Συμφωνία ΓΚΑΤ, συχνά συμφωνούμαστε το γύρο της Ουρουγουάης ως το 92. Όμως η Συμφωνία ΓΚΑΤ επηρεάζει την ΚΑΠ ακόμα και πριν ε, ξεκινήσουν ε, οι δημότες στην Ρουγουάη. Ήδη από τις αρχές τη δεκαετία του 60 με τον γύρο Ντάιλον, όπω έχει ονομαστεί. Και έτσι ξεκίνησαν να εντοπίζονται πολλά προβλήματα καθώ σχεδιαζόταν αυτή η πολιτική, ιδίω με τα υποκατάστατα δημοτριακών και την εισαγωγή ε, προϊόντων σε χαμηλέ τιμέ. Με φυτικέ πρωτενε και αμυλούχα σε χαμηλές τιμές. Το στόχο ήταν να έχουμε φθηνότερα αποκατάστατα δημιουργικών. Όλες οι καταστάσεις για να αποκατασταθεί, να εξορροπηθεί αυτή η κατάσταση, ε, αναχαιτίστηκαν ακριβώς λόγω των κανόνων GATT. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η Συμφωνία GATT δεν επηρέασε την εξέλιξη της ΚΑΠ. Επίσης υπήρχε... Ε, περιορισμένη χρήση των επιστροφών των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Βεβαίω, αυτή τη στιγμή έχει παγώσει στην βαθική κατάψυξη ο γύρο τη Δόχα. Και ο ΠΟΕ δεν θα έλεγε κανεί ότι είναι κινητήρια δύναμη για να οδηγήσει σε μεταρρυθμίσει στην ΚΑΠ. Η τελευταία μεταρρύθμιση του 2013 δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε μεγάλη σχέση με τι διαπραγματεύσει των ΠΟΕ. Και ήταν απλώ μια επαναστάθμιση των προηγούμενων προτεραιοτήτων. Επίση, μου ζητήθηκε να μελετήσω και τι διευρύνσει. Οι διευρύνσει προκάλεσαν αλλαγέ παρά το αγαπημένο όρο του κοινοτικού κεκτημένου υπήρχε νομοθεσία που ίσχυε και συνεχίστηκε να χρησιμοποιεί. Το 1973 όταν ε, προσχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένα θέμα που υπήρχαν πολλά θέματα μάλλον που προέκυψαν ακριβώ λόγω αυτών των διαπραγματεύσεων, όπως οι λιγότερο ευνοημένες περιοχέ ή το τι γινόταν με το Βάμβακα αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος. και την μεταρρύθμιση Φίσλερ μετά τη διεύρυνση του 1996. Ε, όλα αυτά είχαν πολύ σχέση με αυτά που λέγατε. Η διεύρυνση προς την Ανατολική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να σκεφτεί πώς θα συνεχίσει να στηρίζει το εισόδομα των γεωργών με λιγότερο γραφειοκρατικό τρόπο από ό,τι συνέβη με το σύστημα των πρώτερων πληρωμών. Το 2003 έχουμε ήδη ένα πρώτο αποτύπωμα αυτής της ε, τάσης. Νομίζω ότι η διεύρυνση προς τα Ανατολικά λοιπόν έφερε κάποιες αλλαγές στην ΚΑΤ. Είναι ήδη στα σπάργανα οι αλλαγές που σήμερα βλέπουμε να έχουν ολοκληρωθεί. Βεβαίω, όλε οι μείζονε δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που ιδρύθηκε ήταν να δίνει προτιμησιακή πρόσβαση στις ε, απότερες περιοχές, τις υπερπόντιες περιοχές και αυτό ενισχύθηκε μετά την προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ως τάση. Και βεβαίω αυτό διαμόρφωσε την ακροτική πολιτική για την ζάχαρη, τι μπανάνε, το ρύζι και ούτω καθεξή. Επίση, ανελήφθησαν πρωτοβουλίε στα πλαίσια του ΠΟΕ με τι προσπάθειε να βελτιωθεί η ζωή των φτωχότερων χωρών στον κόσμο. Με την ε, πρωτοβουλία λόγου χάρη τα πάντα εκτό από όπλα. Ε, αυτό επηρέασε και το σύστημα εμπορία της Ζάχαρη και ούτω καθεξής. Συνολικά, οι παραχωρήσεις για τα κράτη τη Μεσογείου ήταν λιγότερο γενναιόδορε, βεβαίω. Νομίζω εν μέρη διότι υπάρχουν παραγωγή των ίδιων προϊόντων για την άλλη πλευρά της Μεσογείου και πολλές βρίσκονται σε ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους παραγωγούς της βόρειας ε, πλευράς της Μεσογείου. Εδώ λοιπόν επηρεάστηκε ο τρόπος που καταρτίστηκε η πολιτική στους τομείς αυτούς. Τώρα η έκθεση ολοκληρώθηκε λίγες εβδομάδες ε, πριν με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία. Η προσχώρηση της Τουρκίας δεν μου φαίνεται να είναι μια κοντινή πιθανότητα ε, για το εγγύς μέλλον, όμως εάν υπάρξει τέτοια διεύρυνση, νομίζω ότι οι παραχωρήσεις, οι εμπορικές παραχωρήσεις για τα γεωργικά προϊόντα στην Τουρκία θα δημιουργήσουν πραγματικά προβλήματα στον τομέα της γεωργίας στην Ευρώπη. Αυτό βεβαίω είναι κάτι που για την ώρα δεν πρόκειται να λάβει σε αρκετή από ό,τι φαίνεται. Και επίσης οι πολιτικές γειτονίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωσης δεν ε, ασκούνται μόνο στα νότια αλλά και προς Ανατολέ. Έτσι, οι παραγωγή της Ανατολικής Ευρώπης έχουν βρεθεί στα χαρανάζια της ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία λόγω της στήριξή μας προς την Ουκρανία και μπορεί κανείς να φανταστεί ότι αν αυτού του είδους η ένταση συνεχιστεί και στο μέλλον, εάν η Γεωργία βασίζεται τόσο πολύ στις εξαγωγές, σε δύσκολες αγορές, τότε αν αυτές οι αγορές είναι κλειστές για πολύ καιρό, κάτι θα σημαίνει αυτό. Βεβαίως, με το γύρο της ε, Ντόχας να βρίσκεται στον καταψύκτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες χώρες ανά τον κόσμο προσπαθούν να διαπραγματευτούν νέε ε, συμφωνίες περιοχών ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών. Έτσι, εμεί έχουμε προχωρήσει σε συμφωνίες με την Κορέα. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε σε διαπραγματεύσει μια τέτοια συμφωνία με τον Καναδά, αλλά δεν έχει κυρωθεί. Το πότε θα κυρωθεί, μάλλον το ξέρετε εσεί καλύτερα από ό,τι εγώ ίδιο, με την Μερκοσούρ, την ε, εταιρική σχέση, τη γνωστή διατλαντική συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη ΣΥΠΑ, την TTIP, και ούτω καθεξής. Όπως ξέρουμε για τους Ευρωπαίους γεωργούς, ε, όλες αυτές οι προοπτικές έχουν, ε, ενέχουν μάλλον πολλές προοπτικές, αλλά και κάποιες απειλές λόγω χάρη ε, το κόστος των ε, παρασκευασμένων προϊόντων μπορεί να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε συγκεκριμένε αγορές. Όταν όμως αυτές οι αγορές είναι ιδιαίτερα προστατευμένες όπως η Ιαπωνική ή η Νότιο-Κορεα, νότιο-κορεατική. Βεβαίω υπάρχει όφελο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πετύχει να ειδικέ ειδικε συμφωνία για την πρόσβαση. Όμω άλλε αγορέ όπω τη Αυστραλία και αυτέ θα μπορούσαν να είναι υποφελεί για του παραγωγού τη Ένωση, εάν υπάρχει καλύτερη πρόσβαση για προϊόντα ποιότητα. Βεβαίω η άλλη όψη του ίδιου είναι ότι όταν διαπραγματευόμαστε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με παραγωγούς όπως η Βραζαλία ή η Αυστραλία που παράγουν ε, μαζικά κάποια προϊόντα, τότε βεβαίως ε, οι δικές τους εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι επίσης πολύ Αυτό μπορεί να επηρεάσει ε, τους κτηνοτρόφους και γεωργούς. Αν και ως ακαδημαϊκός και οικονομολόγος πρέπει να πω ότι τελικά οι καταναλωτές αποφελούνται από όλα αυτά. Τώρα, για τις ποσοστώσεις, αυτά μπορούμε κάπως να τα εξορροπήσουμε, να πούμε, ας πούμε ότι η ποσόστοση για το βόλιο θα είναι τόσο ή τόσο. Ε, αλλά σωρευτικά, ο αντίκτυπος των συμφωνιών που συνάπτουμε μπορεί να είναι πιο δραματικός από ό,τι φανταζόμαστε. Ε, λόγω χάρη, αν υπάρξει μια συμφωνία ελεύθερων ε, εμπορικών συναλλαγών με όλες τις χώρες του κόσμου, και περιορισμό των δασμών ε, σε επίπεδο ΠΟΕ, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Όμω, έτσι αλλιώ πρόκειται να εκδώσει έκθεση κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του θέματος. Να περάσω τώρα από τα εμπορικά ζητήματα για λίγο σε κάτι άλλο. Η προσφατότερη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, όπως είπα, έγινε το 2013. Ένα από τα βασικότερα στοιχεία τη ήταν το στοιχείο του πρασινίσματο, το οποίο μεταξύ άλλων ε, είχε να κάνει με την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τι γεωργικές δραστηριότητε. Αυτή τη στιγμή είμαι και εγώ στο στρατόπεδο των σκεπτικιστών σε αυτή την παράταξη. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι τα μέτρα που προτείνονται και έχουν εγκριθεί θα το πετύχουν αυτό με τρόπο που θα είναι και αρκετά οικονομικό. Κοιτάζω τα στοιχεία που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τα κοιτάζω την ερχόμενη διετία για να δούμε κατά πόσο είναι πολιτικέ μα είναι αποτελεσματικέ. Όμω έχω την εντύπωση ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μάλλον ο κόσμο, για να είμαι πιο σωστό, θέλει να πετύχει τι προσδοκίε τη παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα, θα πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί πιο αποτελεσματική για τη μείωση του ενέργειου του θερμοκηπίου. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και μετά το διάστημα του 2020 και τον περίοδο μετά το 2020 για την ΚΑΠ. Σύντομα συμπεράσματα. Ποια είναι τα ζητήματα, ε, τα, ποια είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι που επηρεάζεται από τις εξωτερικές εξελίξεις τελικά. Όμως δεν νομίζω ότι ο ΠΟΕ θα επηρεάσει πάρα πολύ το τι θα συμβεί στην ΚΑΠ μέχρι το 2020. Μετά την πρόσφατη μεταρρύθμιση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη για άμεσες αλλαγές. Μάλιστα, ήταν πιο επικίνδυνο να έχουμε περιβαλλοντικά προγράμματα που δεν είχαν να κάνουν πάρα πολύ σχέση με το πράσινο κουτί, αλλά περισσότερο με το κίτρινο, γιατί θεωρείται ότι εκεί ήταν πιο ταιριαστά. Αυτό δεν ξέρω αν έφερε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Επίση, θα χρειαστεί ένα καλύτερο μηχανισμό επίλυση διαφορών για το μέλλον, αρκεί να το θέλουμε. Ένα συγκεκριμένο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι οι κανόνε του πρασινίσματο πρέπει να αναθεωρηθούν για να βεβαιωθούμε ότι η Γεωργία όντω μειώνει τι εκπομπέ αερίου του θερμοκηπίου. Και ένα τελικό σχόλιο, αν με επιτρέπετε, για το Brexit. Νομίζω αυτό θα σημάνει μάλλον ότι θα έχετε λιγότερα κονδύλια για τον πλογισμό τη γεωργική πολιτική για μετά το 2020, αναλόγω με το αποτέλεσμα των διαμαρτύρων. Όμω, ό,τι συμφωνία και αν πετύχουμε ε, για μα και του ε, Βρετανού, θα επηρεαστούν σίγουρα οι ροέ γεωργικών προϊόντων ή η Ιρλανδική κτηνοτροφία, που θα αντιμετωπίσει αρκετέ διακυμάνσει και τριγμούς λόγω του Brexit. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε που με επιτρέψατε να κάνω αυτή την σύντομη παρουσίαση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Περνάμε στη συζήτηση. Ερωτήσεις και σχόλια των Ευρωβουλευτών. Και μετά θα σας ξαναδώσουμε το λόγο, κύριε Σουίμπανκ. Ο κύριος Φλάνναγκαν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Όσον αφορά τις εξωτερικές πιέσεις, οι γεωργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφερθήκατε στους κτηνοτρόφους της Ιρλανδίας ε, ανακουφίστηκαν όταν ε, ο Φιλ Χόγκαν είπε τον ε, Μάιο ότι το μοσχαρίσιο κρέας δεν βρίσκεται πλέον ε, πάνω στο τραπέζι. Ότι έχει ε, αφαιρεθεί από τις συμφωνίες με τις χώρες της Mercosur. Είναι ε, ρεαλιστικό να περιμένουμε οι χώρες της Μερκοσούρ να καταλήξουν σε σύναυση συμφωνίας που δεν θα περιλαμβάνει το βόηο κρέας. Αυτό είναι μια εξωτερική πίεση που εμείς δεν την περιμέναμε. Ποια είναι η δική σας γνώμη για αυτό το θέμα και θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Γιατί ε, είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ως θέμα συζήτησης και τελικά βλέπουμε τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο κύριος Άγνιο. Ο κύριος Φλανάγκαλ έκανε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο. Το Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω είπε ότι βγήκε από το μενού το βοδινό αλλά αυτό ίσως ε, ε, θα ενθάρρυνε στους Βρετανούς αγρότες ε, να ψηφίσουν υπέρ παραμονής, γιατί φοβούνταν μήπω κατακλειστούν από το Μερκόσουν και καθυσυχάστηκαν με αυτή τη διαβεβαίωση. Βέβαια τώρα με τον Brexit πάλι εντάθηκαν οι ανησυχίες. Ό,τι αφορά τις δραστηριότητες της ΕΙΕΔ και την κοινή γεωρική πολιτική. Όπω είπε και ο πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν τεράστια προβλήματα ε, και που δημιουργήθηκαν με το ρωσικό εμπάργο για τη ευρωπαϊκή γεωργία και αρνητικό αντίκτυπο ε, είχαμε αντιμετωπίσει και εμείς τα προβλήματα. Ήμουν στην αρχή της εβδομάδας ε, στην Ιρλανδία. Ήλπιζα να δω και τον κύριο Φλάναγκαν, αλλά απουσίαζε. Μάλλον δεν άντεχε ούτε ζωγραφιστό να δει τον κύριο Φιλ Χόγκαν. Ε, πάντως εντυπωσιάστηκα από το πώς ε, ε, οι, οι αγρότες θέλουν να ελέγξουν τον καιρό. Κάποια με γιουχάησαν, αλλά τελικά ε, ήρθε κάποιος και με συνεχάρη, γιατί φαίνεται ότι ε, κατάλαβε το σχολείο μου για το πόσο ε, θα εμποδιστούν οι, οι γεωργοί όταν ε, σταματήσουν οι αγελάδες να κάνουν κάτι που φυσικά πρέπει να κάνουν προσπαθώντας να μειώσουν τη συμμετοχή τους στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου. Μάλιστα συνάντησε και ένα νεαρό γεωργό από τη Σλοβενία και μου είπε ότι πολλοί από τους συμπατριώτες τους αγοράζουν τώρα χωράφια στη Σερβία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν επιβάλλονται κυρώσει ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των σερβικών προϊόντων. Και κάτι τέτοιο στηρίζει και αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το μήνυμά μου προ την ΙΕΔ είναι ότι δημιουργείται πολλά προβλήματα μόνο, αλλά απολύσει τίποτα. Η ε, κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το τμήμα πολιτικής για την έκθεση, γιατί είναι σημαντικό να δούμε τη, τον αντίκτυπο που έχει η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινή γεωργική πολιτική. Μια και έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα σταθώ σε έλεγα σημεία. Είπατε ότι δίνει ευκαιρίες και συμφωνώ μαζί σας, κυρίως σε προϊόντα ποιότητας, εξασφαλίζει πρόσβαση σε αγορές με αντίστοιχες προδιαγραφές και με αντίστοιχο βιωτικό επίπεδο με το δικό μας. Μπορεί να δίνει ευκαιρίες για τέτοιου είδους προϊόντα. Αλλά έχουμε ταυτόχρονα και απειλές ε, αναφυσβήτητες. Είπατε ότι όταν συνάπτουμε συμφωνίες ε, με χώρες ε, παρόμοιες με μας, με αντίστοιχες προδιαγραφές και με παρόμοιες τιμές, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και αποφελούνται οι καταναλωτές. Βγαίνουν κερδισμένοι οι καταναλωτές δηλαδή όταν μειώνονται οι τιμές. Δεν συμφωνώ με τη διαπίστωση αυτή, γιατί θεωρώ ότι αν έχουμε από την αρχή τον ανταγωνισμό μόνο σε επίπεδο τιμών και μία κούρσα για τη μείωση των τιμών ε, υπέρ των καταναλωτών, σε τελική ανάλυση δεν θα υποφεληθούν οι καταναλωτές ε, από χαμηλές τιμές, γιατί θα επιδεινωθεί τόσο η κατάσταση του κλάδου που θα είναι αντιπαραγωγικό. Οπότε ε, η ανταγωνιστικότητα των συμφωνιών ε, με επιρροή στην μείωση των τιμών είναι κάτι θετικό για τους καταναλωτές. Μπορεί αυτό να ισχύει, αλλά μόνο σε αρχικό στάδιο. Μετά ανατρέπεται. Επίσης, ε, δημιουργούμε τεράστιες πιέσεις και ανταγωνιστικές πιέσεις στην ποιοτική παραγωγή που είναι πολύ υψηλή, υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, δεν θα πρέπει να τις υποβαθμίζουμε με μια ανταγωνιστικότητα που επικεντρώνεται μόνο στις τιμές. Επίσης, αυτό που με προβληματίζει είναι η έλλειψη αμοιβαιότητας στις συμφωνίες. Όταν δεν έχουμε αμοιβαιότητα και στις προδιαγραφές και στα πρότυπα και παρόλα αυτά συνάπτουμε εμπορική συμφωνία, τι συμβαίνει, αποδυναμώνεται ο Ευρωπαίος Γεωργός και η δική μας επιστηστική βιομηχανία. Γιατί εμείς έχουμε υψηλές προδιαγραφές ε, και δεν τηρούνται από όλους και στη τελική ανάλυση καταναλωτές καταναλώνουν προϊόντα από άλλες χώρες, ε, ντομάτες από το Μαρόκο ε, και τα αντικαθιστούν με τέτοια προϊόντα εισαγόμενα τα απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να κάνει μερικές φορές μια εμπορική συμφωνία. Βέβαια δεν ισχύει πάντα αυτό. Οπότε η αμοιβαιότητα είναι ουσιώδες στοιχείο και διαφοροποιητικό των συμφωνιών. Μόνο συμφωνίε με αμοιβαιότητα θα κάνουν τη διαφορά. Και επίση, ε, δεν ξέρω τι ε, επιπτώσεις θα έχει το greening. Πάντως προ το παρόν ε, μου φαίνεται μόνο ω γραφειοκρατικό κατασκεύασμα και θα πρέπει να διορθωθεί. Και θα πρέπει να διορθωθεί χάρη στι προτάσεις απλούστευσης. Είμαι υπέρ ε, του πρασινίσματος Τη οικολογικοποίηση, αλλά πολύ αμφιβάλλον η παρούσα πρόταση για το greening θα μας εξασφαλίσει ένα τέτοιο πιο περιβαλλοντικό χαρακτήρα της γεωργίας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κούσμιακ, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την εκπόνηση αυτής της μελέτης, που είναι ένα παύγασμα γνώσεων ε, για τις αλληλεπιδράσεις ε, της εξωτερικής πολιτικής στη γεωργική πολιτική πολύ ενδιαφέρον το πώς επηρεάζουν οι εξωτερικές μας δράσεις στην γεωργική μας πολιτική. Έχω δύο ερωτήσει προς τον εμπειρογνώμονα, τον κύριο καθηγητή. Είναι αναφυσβήτητο ότι το άνοιγμα της ενωσιακής αγοράς σε προϊόντα τρίτων χωρών με την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών ε, κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο γιατί πολλές διαπραγματεύσεις διεξάγονται ταυτόχρονα αλλά πολλές φορές οι συμφωνίες αυτές αφορούν χώρες που δεν είναι σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση που τηρεί ψηλέ προδιαγραφές για την καλή μεταχείριση των ζώων, την ευζοία, την οικολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις κλιματικές αλλαγές. Μερικές χώρες επικεντρώνονται μόνο στο κόστος παραγωγής. Οπότε, πώς μπορούμε να προασπίσουμε τη γεωργία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τέτοιου είδους αθέμητο ανταγωνισμό από χώρες που ε, έχουν χαμηλές προδιαγραφές. Σε ό,τι αφορά το Brexit, είπατε ότι το Brexit θα έχει χαμηλότερη επίδραση στην ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία και λιγότερη επιζήμια από ότι το ρωσικό εμπάργο. Ε, παρά είναι σοβαρή αυτή η διατύπωση, αλλά για το ρωσικό εμπάργο ε, χρειάστηκαν περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε τις επιμέρους γεωρικές αγορές. Γι' αυτό και είναι πολύ ζωφερή αυτή η προπτική για τις επιρροές που θα έχει ενδεχομένω και το Brexit στις γεωργικές αγορές. Ο κύριος Χόισλινγκ. Πιστεύω ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να συζητήσουμε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα του ΚΟΡΚ. πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, γιατί ακούγονται διάφορες ε, απόψεις. Ιστορικά, η εξέλιξη του δεύτερου πυλώνα ήταν το αποφασιστικό βήμα για τον εξυγχρονισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής. θα κάνουμε λοιπόν απροηγόθετες πληρωμές ε, στον πρώτο πυλώνα ή θα δώσουμε περισσότερο χώρο, χώρο στο δεύτερο πυλώνα, στο μέλλον. Είπατε ότι το ελεύθερο εμπόριο, αυτό αυτό ωφελεί τους καταναλωτές και ότι θα πρέπει από αυτή την άποψη να επιδιώξουμε να συναφθούν ε, αντίστοιχες συμφωνίες και με την Αυστραλία και με άλλες χώρες. Ε, εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώ έτσι. Μπορεί βραχυπρόθεσμα να εμφανίζονται κάποια ωφέλη, αλλά το να εκθέσουμε τις δικές μας επιχειρήσεις και την οικονομία μας σε ανταγωνισμό με τις Αυστραλιανές ή με τις Αμερικάνικες επιχειρήσεις, νομίζω ότι θα δημιουργήσει πολύ, μεγάλες, πολύ μεγάλα προβλήματα και πολύ μεγάλες δυσκολίες ε, στην ε, Ευρώπη. Εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις δομές των ΙΠΑ έτσι απλά και να πούμε ότι καταργούμε όλα τα εμπόδια και το μόνο που μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα είναι η ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών. Αν θέλουμε δηλαδή να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Γεωργία, κάτι που θα ωφελήσει μακροπρόθεσμα και τους καταναλωτές, τότε νομίζω ότι θα πρέπει σε έναν μικρό βαθμό τουλάχιστον να υπάρχει και μια εξωτερική προστασία. Και νομίζω ότι θα ήταν μοιραίο είναι μοιραίο το γεγονός ότι ο ε, Επίτροπος σε όλα τα διεθνή φόρα ε, προσπαθεί να ανα, ανοίξουν οι άλλες χώρες τις αγορές τους. Μα και οι άλλες χώρες αυτό θα απαιτήσουν από εμάς, αν το απαιτούμε εμείς. Γι' αυτό ε, νομίζω ότι το κυριότερο για μας δεν είναι μόνο να ασκούμε μια επιθετική εξωτερική πολιτική, επιθετική ως προς τις εξαγωγές ενώ ε, Αντιθέτως νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και πολλές άλλες διαστάσεις. Είπατε ότι ο γύρος της Ντόχα έχει πεθάνει στην ουσία. Άρα δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν θα πρέπει και εμείς να προστατεύσουμε τις δικές μας αγορές ε, από τον διεθνή ανταγωνισμό. Ακριβώς γιατί θέλουμε να ε, διατηρήσουμε και την ε, ευρωπαϊκή γεωργία και τις δικές μας μεθόδους ε, καλλιέργειας και εκτροφής. Όσον αφορά αυτά που είπατε για τη Συμφωνία των Παρισίων, για το κλίμα, εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους εκείνης της συμφωνίας μέσω ορισμένων ε, απλών διατάξεων για το πρασίνισμα. Νομίζω ότι θα απαιτηθεί μια πολύ ε, βαθύτερη συζήτηση για να επιτύχουμε, επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ. Καταρχήν ε, να πω ότι ονομάζομαι η Μακουλάτ Πινιέρο, είμαι μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Γεωργίας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ πάντως για την παραγγελία αυτή τη ε, μελέτη που είναι πολύ σημαντική και καλό είναι να εγγύψουμε σε αυτά τα θέματα από κοινού και να ευχαριστήσω τον ε, συντάκτη της μελέτης αυτής ε, για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλιά του. Έχω μια ερώτηση ε, και θα ήθελα και τη γνώμη της Επιτροπής σας, αν επιτρέπει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής Γεωργίας για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ό,τι αφορά το άνοιγμα και άλλων αγορών ή το συντονισμό ε, στο, στα φυτογειονομικά θέματα και τις ε, φυτογειονομικές ε, νομοθετικές διατάξεις, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους Γιώργους. Και αυτό που λείπει είναι οι αλληλεπιδράσεις με την πολιτική της αναπτυξιακής συνεργασίας. Γιατί ε, η Ευρωπαϊκή Γεωργία είναι πολύ σημαντική γιατί την υπερασπίζομαι με νύχια και με δόντια και συμφωνώ με την κυρία Γκυλέρο, θα πρέπει να ισχύουν συνθήκες ε, θεμητού ανταγωνισμού. Όταν όμω έχω, ασκούμε εμπορική πολιτική και κυρίω με τρίτε χώρε λιγότερο αναπτυγμένες, συσχετίζουμε τι εμπορικέ μα συμφωνίε με την αναπτυξιακή μα βοήθεια και συνεργασία και διευκολύνουμε αυτέ τι χώρε να διαθέτουν τα προϊόντα του στη δική μα αγορά. Βέβαια τώρα έχουν εξειδικευμένε παραγωγέ, θέλουμε να του βοηθήσουμε να διαφοροποιήσουν την οικονομία του. Οπότε αυτό θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε την αλληλεπίδραση γεωργικής και εμπορικής πολιτικής. Επίσης, ε, θα ήθελα να μάθω από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γνώμη έχει σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Γιλέρα. Η κυρία Γιλέρα είπε ότι επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωρικών Προϊόντων ε, παρόλο που αυτά δεν υπόκειται στους ελέγχους και τις υψηλές προδιαγραφές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως και ένα επιπλέον πρόβλημα. Στα λιμάνια μας ε, φτάνουν προϊόντα και στα σύνορά μας φτάνουν προϊόντα και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει συντονισμένη πολιτική, φορολογική και ελέγχου της ποιότητας στα τελωνία, περνάνε ανεξέλεγκτα προϊόντα από τα σύνορά μας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το παραμελήσουμε. Θέλουμε μια εναρμονισμένη πολιτική απαιτήσεων, προδιαγραφών και με τους κατάλληλους πόρους για να γίνονται καλύτερη επιθεωρήσεις και η έλεγχη των εισαγόμενων προϊόντων. Γιατί είχα θέσει αυτή την ερώτηση και μου απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Πιστεύετε πραγματικά ότι δεν χρειάζεται να μεριμνήσουμε ώστε όλα τα προϊόντα που φτάνουν στην Ευρώπη να πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τους Ευρωπαίους Γεωργούς, γιατί αν γίνει δυνατό κάτι τέτοιο, έρχονται σε πολύ δυσμενή θέση, σε αθέμητο ανταγωνισμό και έτσι έχουμε απώλεια των προδιαγραφών ε, κατανάλωσης και ποιότητα που ισχύουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξαιτία αυτού του ανταγωνισμού υποβαθμίζονται. Σας ευχαριστούμε κύριε Πινιέρο για την παρουσία σας καταρχήν και για τα σχόλιά σας. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερος ε, όταν και άλλες επιτροπές ασχολούνται με γεωργικά θέματα. Η Επιτροπή Εμπορίου, η Επιτροπή Εξωτερικών, η Επιτροπή Ανάπτυξης και ενθαρρύνουμε τις υπόλοιπες επιτροπές να ασχολούνται με γεωργικά θέματα γιατί μας ε, θλίβει όταν οι υπόλοιπες επιτροπές ε, περιορίζουν το δικαίωμά μας ε, να διευρύνουμε τον προβληματισμό μας. Γιατί η Επιτροπή ΑΦΕΤ και η Επιτροπή Εμπορίου μπλόκαραν την πρότασή μας για έκθεση των εξωτερικών πτυχών και παραγόντων που, επηρεάζουν την γεωρική πολιτική. Ενώ εμείς θεωρούμε ότι έχουμε δικαίωμα να ασχολούμαστε με τις εξωτερικές πτυχές, παρόλο που μερικοί θεωρούν ότι έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο. Εμείς ξέρουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας, ξέρουμε ότι θέλετε συντονισμό, αλλά ακούστε και τη δική μας γνώμη. Και γι' αυτό είχαμε ε, σύγκρουση αρμοδιότητων με δύο επιτροπές και τελικά αλλάξαμε τη διατύπωση και δώσαμε αυτή την μορφή τελικά στην έκθεση προκειμένου να μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε προς τις άλλες επιτροπές. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερω για την παρουσία σας ε, και ελπίζω τα σχόλιά μας να τα διαβιβάσετε και στην Επιτροπή στην οποία είστε μέλος, στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος επίσης ε, εξετάζονται μερικά γεωργικά θέματα και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Και είναι σημαντικό να παρουσιάζουμε με θετικό φως τα γεωργικά θέματα και στις άλλες επιτροπές. Ε, λυπούμε που έκανα αυτό το σχόλιο, αλλά το θεώρησα σκόπιμο αυτή τη στιγμή. Η κυρία Ντελέ κυρία Ντελέ που θα είναι και η συγγήτρια τη σχετική έκθεση, που επαναλαμβάνω χρειάστηκε να τροποποιήσουμε κάπω τον τίτλο και το περιεχόμενο. Και να του δώσουμε τη μορφή που είχε και η μελέτη που ζητήσαμε από το Γραφείο Πολιτικών. κυρία Ντελέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δείξατε το καθοριστικό θέμα από το όλο αυτό ζήτημα. Η ευρωπαϊκή γεωργία και το μέλλον της στον κόσμο είναι κάτι που σε κάθε χώρα απασχολεί τους γεωργούς και μας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την παρουσίαση. Υποδείξατε τη σημασία και την επίδραση των εξωτερικών εξελίξεων στην ΚΑΠ. Κάποιες φορές η επιρροή ήταν θετική, αλλά θεωρώ ότι υπήρξαν και αρνητικές πτυχές συνέπειες επιβλαβής για, ορισμένους, για ορισμένες αποφάσεις που ελήφθησαν. και για μια σειρά από συμφωνίες ε, τις οποίες ε, ήδη έχουμε συνάψει είπε η κυρία Αγγιλέρα τι γίνεται με τις ντομάτες από το Μαρόκο ή που βρισκόμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων. Η γαλλική, ισπανική, η ιταλική παραγωγή έχουν πληγεί από την συμφωνία με το Μαρόκο λόγω και το ρελόδο με την είναι κάτι παρόμοιο. Ξέρετε πόσο οι συνέπειε δεν έχουν τον ίδιο τύπο παντού. Εδώ λοιπόν για μένα είναι ζήτημα αρχής και τρόπου με τον οποίο θα λειτουργούμε. Ο κίνδυνο αυτός υπάρχει και για το βόλιο κρέα με την Μερκοσούρ με το TTIP αλλά και με τη συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά, νομίζω ότι πρέπει να ε, γίνει μια ε, ανάπαυλα, όπως υπόθηκε σε μια ακρόαση, ως προς τα ζητήματα αυτά. Πρόεδρε, ε, είπατε είμαστε υποχρεωμένοι να μελετήσουμε το θέμα από μια άλλη οπτική γωνία. Μου φαίνεται καθοριστική σημασία. Διότι η παρουσίαση καταλήγει στην, στο εξή συμπέρασμα. Όλα αυτά εντείνουν την εκείμανση των τιμών στην αγορά γεωργικών προϊόντων. Οπότε, προδήλω, και το σημειώνουμε με ιδιαίτερη ε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ε, με οξυμένο ενδιαφέρον λόγω του ρωσικού εμπάργου, τα θέματα αυτά, οι αυτές έχουν ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπατε, διεξαγάγει εξωτερικέ πολιτικέ που είναι και προ όφελο των Ευρωπαίων Γεωργών και εκτροτρόφων. Το θέμα τη διακύμανση των τιμών βρίσκεται στο κέντρο αυτών των μεριμνών και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να ισχύει αυτό και για την επόμενη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τον εμπειρογνώμονα για την παρουσίασή του. Πώς συνδέονται λοιπόν η γεωργική με την εξωτερική πολιτική. Δεν πιστεύετε κι εσείς ότι το όλο θέμα σχετίζεται και με το θέμα του εμπάργου κατά της Ρωσίας και ότι ε, υπάρχει μια κάποια ε, έλλειψη αξιοπιστίας στο όλο θέμα. Για παράδειγμα, στα διαστημικά θέματα συνεργαζόμαστε μια χαρά με τη Ρωσία στα γεωργικά πάλι τους επιβάλλουμε εμπάργο. Και ε, αυτός που έχει πληγεί περισσότερο από όλους ε, από το εμπάργο αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Γεωργία Ελπίζω λοιπόν να σταματήσει γρήγορα το εμπάργο αυτό. Είπατε για τον ΠΟΕ, για το γύρο της Ντόχα και τα λεφτά. Μήπως θα ήταν καλύτερο να αναζωογονθεί, να ανασυσταθεί αυτός ο γύρος της Ντόχα παρά να συνάπτουμε επιμέρους συμβάσεις διμερείς ε, ελεύθερων εμπορικών ε, συναλλαγών όπως με τη Μερκοσούρ ή το TTIP. Εγώ λυπούμαι που δεν υπάρχει πια αυτός ο γύρος της ε, Ντόχα. Όσον αφορά το ελεύθερο εμπόριο και τις σχετικές συμφωνίες, και εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν ε, ευκαιρίες αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι. Αναφερθήκατε στο θέμα του βόηου κρέατος. Εσείς πιστεύετε ότι σε περίπτωση που συναυθούν τέτοιου είδους ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου δεν θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ανώτατα όρια για τις εισαγωγές στο βόηο κρέας για παράδειγμα. Είπατε και για το πρασίνισμα. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα διάβασα μια έκθεση από την Βαβάρια όπου αναφέρεται ότι τα σχετικά μέτρα για το πρασίνισμα ε, είχαν μέχρι στιγμής ε, θετικό αντίκτυπο στην ε, γεωργία. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε πολλούς τομείς Παρόλα αυτά πρέπει να πούμε ότι τα, οι διατάξει για το πρασίνισμα θα ήταν ακόμη πιο αποτελεσματικές αν δεν συνοδεύονταν από γραφειοκρατικές ε, διαδικασίες που επιβάλλουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Θέλω να πω ότι οι γεωργοί έχουν φτάσει πλέον στο σημείο να λένε ότι δεν θέλουμε οι εθνικές κυβερνήσεις να θεσπίζουν κανόνες για αυτά τα θέματα, ρυθμίστε τα εσείς από τις Βρυξέλλες. Μήπως τελικά ε, είναι καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις να θεσπίζετε ευρωπαϊκή νομοθεσία και να μην, αφήνετε, να μην αφήνονται τα θέματα αυτά στις εθνικές κυβερνήσεις. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο από την Επίτροπο Ίντα, από την Επιτροπή Ίντα, Εγώ ε, ήμουν για πολλά χρόνια μέλος αυτής της Επιτροπής. Δυστυχώς αυτή τη φορά, σε αυτή τη θητεία δεν τα κατάφερα να γίνω μέλος της γιατί δεν υπήρχαν ε, διαθέσιμες θέσεις. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ε, συμφωνήσω μαζί σας ότι στις διαπραγματεύσεις για τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει εμείς να επιμένουμε στις δικές μας, στην τήρηση των δικών μας προδιαγραφών. Το 2010 σε έκθεσή μου είχα ε, προτείνει ε, να επιτρέπονται οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων μόνο εφόσον τηρούνται οι ευρωπαϊκές ε, προδιαγραφές για το περιβάλλον, για την εκτροφή, για την καλλιέργεια κτλ. Μάλιστα, η έκθεσή μου αυτή είχε υπερψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία, με 534 ψήφους στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Αυτά ε, ήθελα να πω από την πλευρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πετήρ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον καλεσμένο μας για την πολύ αξιόλογη παρουσίαση τη μελέτης. Όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, στην Γεωργία είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών αποφάσεων, όπως είπατε και εσείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει στο μέλλον ε, να, είναι πιο σταθμισμένη, γιατί ε, δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη τις ε, επιπτώσεις που θα έχει στη συνέχεια στη, στους γεωργούς μας και στη γεωργία. Η Κροατία έχει μια ασταθή και ευάλωτη αγορά και βρίσκεται υπό τεράστιες πιέσει, όχι μόνο το, από τρίτες χώρες, πιέσεις και από τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και συμφωνώ ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις νέες δημοκρατίες στι τρίτε χώρε, να τις βοηθήσουμε στο δημοκρατικό τους δρόμο, αλλά όχι εις βάρος των δικών μας, των Ευρωπαίων ε, Γεωργών. Δεν ξέρω ποια είναι η πρότασή σας για να αντισταθμίσουμε τις επιζήμιες συνέπειες της εξωτερικής μας πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Γεωργία ή τι προστατευτικά μέτρα θα μπορούσαμε να λάβουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τους γεωργούς μας από τον αθέμητο ανταγωνισμό. Και έχω και μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, ε, όπως και η Κροατία, εισάγουν ε, ε απορροκυπευτικά από τρίτες χώρες. Μάλιστα απορροκυπευτικά που ε, υπόκεινται σε χημικές επεξεργασίες από δραστικές ουσίες που απαγορεύονται στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εμείς χρησιμοποιούμε, εισάγουμε προϊόντα που, ε, στα οποία έχουν εφαρμοστεί ζανιακτόνα και φυτοκτόνα που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός κατά των Ευρωπαίων γεωργών. Βέβαια είναι πιο φθηνά αυτά τα προϊόντα, αλλά είναι επιβλαβή για την υγεία των καταναλωτών. Και επιπλέον, επαναλαμβάνω, συνιστούν αθέμητο ανταγωνισμό για τα ευρωπαϊκά προϊόντα που πληρούν τις υψηλέ ε, ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ε, θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα κατά αυτών των προϊόντων. Τι προστατευτικά μέτρα σκοπεύετε, δίνονται ε, να λάβουν τα κράτη-μέλη για να αποτρέψουν την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων που έχουν ε, παραχθεί με φυτογεωνομικά μέτρα ή προϊόντα φάρμα, ε, ζανιοκτώνα που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπογκόβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτή τη μελέτη, η οποία ήταν εξαιρετική και στην παρουσίασή σας και νομίζω ότι τα πήγατε πολύ καλά για να μας εξηγήσετε πώς η Ευρωπαϊκή Γεωργία και η πολιτική της είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εξωτερική πολιτική και τις εξωτερικές εξελίξεις. Το είδαμε αυτό πρόσφατα σε γεγονότα όπως η κατάρριξη των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, το ρωσικό εμπάργκο. Είδαμε πως τα ακόμη και τα πιο πρόσφατα γεγονότα μπορεί να έχουν επίπτωση στην ΚΑΠ. Δεν θέλω να σχολιάζω την κατάσταση με τη Ρωσία, αλλά το τίμημα φαίνεται να το πληρώνουν οι γεωργοί. Την διαμάχη αυτή Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Ελπίζω ότι οι επιπτώσεις θα είναι μόνο βραχυπρόθεσμες. Όμως, στο μεταξύ, ο ρωσικός κοινωνικός τομέας προσαρμόζεται. Ένα ευρωπαϊκός θα πρέπει να επιφέρει σοβαρές αλλαγές για να τα καταφέρει. θα πρέπει να μην καταλήξουν οι Ευρωπαίοι Γεωργοί να είναι πιόνια στη σκακέρα των διεθνών διπλωματικών σχέσεων. Επίσης, να μην ξεχνάμε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εμπορικές σχέσεις έχουν τεράστιες επιπτώσει στην παραγωγή τροφίμων. όπως είπε και η κυρία Πετήρα από την Κροατία, πρέπει να προσέξουμε να μην βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ισοπεδωμένο σύνολο, η Γεωργία για ανάγκες της και τα χαρακτηριστικά τους, και τα χαρακτηριστικά της είναι πολύ διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Η τάδε εμπορική συμφωνία, λόγου χάρη, μπορεί να είναι πολύ πιο αρεστή σε αυτούς που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί από ότι σε αυτούς που δεν είναι. Πρέπει να προσέξουμε, να βεβαιωθούμε ότι οι αρχές της ΚΑΠ συνεχίζουν να ισχύουν και ότι παράγονται μεν σωστέ ποσότητε, αλλά γι' αυτό έχουν και το κατάλληλο εισόδημα, την κατάλληλη αμοιβή οι γεωργοί. Δηλαδή λαμβάνουν ε, τι τιμέ που αξίζει η παραγωγή των προϊόντων του, σεβόμενοι ταυτόχρονα το περιβάλλον. Αυτά τα διάφορα στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη ταυτόχρονα. Σε καιρού όπω η τωρινή που είναι σχετικά δύσκολη, ε, που οι αλλαγέ είναι πιο δύσκολο να μεταφερθούν, που έχουμε την ε, συμφωνία ΣΕΤΑ ε, με τον Καναδά σε συζήτηση, ξέρουμε ότι είναι σαν να κάνουμε ένα άλμα στο κενό έχουμε ξεπεράσει τα ε, όρια που πρέπει για να προτεύουμε τους Γιωργούς ή όχι. Ο κύριος Δεκάστρο, ευχαριστώ κύριε καθηγητά για τη μελέτη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, αλλά τόνισαν και πολλοί συνάδελφοι, η ΚΑΤ πληρώνει πολλές φορές ε, τις συνέπειες των ε, εξωτερικών επιλογών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέπειες πολλές φορές οφείλονται στο ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αμοιβαιότητας όπως θύμασε και η συνάδελφος Αγγιλέρα αλλά να ευχαριστήσω και την Εμακουλάδα για την διαπίστωση που έκανε, για την παρατήρηση που έκανε. Ε, πρόεδρε, θέλω να μιλήσω τώρα για το εξή. Ε, συχνά μιλάμε για την επιρροή, δυστυχώ το επισημαίνω γιατί μα αφορά και εμά άμεσα, για τι συνέπειε τη εξωτερική πολιτική στην ΚΑΠ. Δεν θα πρέπει όμω να φωτίσουμε για τι συνέπειε που μπορεί η ΚΑΠ να έχει στην εξωτερική πολιτική τη Ένωση. Αντιστρόφω δηλαδή. Ε, πόσο ενδιαφέρον θα ήταν να δούμε τι τις εμπειρίες που είχαμε από την Ευρώπη με τις πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου τα προγράμματα LEADER. Δηλαδή κάθε φορά ε, που θέλουμε να ξεκινήσουμε μια νέα πρωτοβουλία και περνάμε σε συνεργασία με χώρες της Βορειάς Αφρικής, το Μαρόκο, την Τινησία, το μόνο που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να ανοίγει τα σύνορα της Ένωσης, κάθε φορές και, κάποιες φορές και λίγο αληθορίζοντας, όχι πάντοτε με τον ίδιο τρόπο, δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο τα κράτη βορείως και νοτίως της Ευρώπης. Όμως θα μπορούσαμε να είμαστε θετικοί. Προγράμματα ανάπτυξης υπαίθρου θα μπορούσαμε να προτείνουμε και στις χώρες αυτές, να τα εξάγουμε, όταν υπάρξει ευρωπαϊκή στήριξη στήριξη ε, από τα χαμηλά. Να ξαναπιάσουμε τη στήριξη των χωρών αυτών που έχουμε εγκαταλείψει, να προτείνουμε προγράμματα ανάπτυξη πέθρου αυτού ε, με ευρωπαϊκή δομή. Τα οποία να τα αναλάβουν στο τοπικό επίπεδο. Αυτό θα αντέστρεφε κάπω τι σημερινέ τάσει. Επίση, να δούμε πω η ΚΑΠ μπορεί να επηρεάσει θετικά τι εξωτερικέ ε, δράσει τη Ένωση με τέτοιε πρωτοβουλίε συνεργασία που δεν θα ε, περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο σε μια ανταγωνιστική σχέση για την θέση σε αγορά συγκεκριμένων προϊόντων, αλλά με μια προσπάθεια σοβαρή, ε, ειλικρινή, για να προωθήσουμε τη γεωργία σε αυτέ τις χώρες, ίσως και αξιοποιώντα αυτού του ίδιου του κανόνε τη ΚΑΠ. Ευχαριστούμε κύριος Νίκολσον. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Σουίνμπαν για την παρουσίασή σας. Η αλήθεια είναι, είναι ότι αν κοιτάξει κανείς όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσει του ΠΟΕ, τη ΤΕΤΗ, με τη Μερκοσούρ, την Αυστραλία, την Αζηλανδία και το καθεξής, θα δείτε ότι υπάρχουν θέσεις ε, επιθετικές και αμυντικές. Θα πρέπει λοιπόν κανεί να αποφασίσει αν θα έχει εμπορικέ διαπραγματεύσει ή αν θα περάσει στον απομονωτισμό. Πρέπει κανεί να αποφασίσει τι γραμμή θα τηρήσει. Η αλήθεια είναι. Και αναφέρατε τι γίνεται με τις τιμές εισαγωγέ από άλλε χώρε. Εγώ ήμουν μέλος τη επιτροπή αυτή σε μια επίσκεψη ε, στη Βραζιλία, όταν πήγαμε μια επίσκεψη στη Βραζιλία, τη στιγμή που υπήρχε όλο αυτό το θέμα με το βραζιλιάνικο βόλιο. Ε, Μα είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα, η Βραζιλία ανταποκρίνεται στα πρότυπα παραγωγή του βόλου. Ήταν άλλο ο πρόεδρο τότε τη Επιτροπή μα ε, και δεν ε, είχε καθόλου δίκιο η Επιτροπή, διαπιστώσαμε όταν πήγαμε εμείς στη Βραζιλία, με αυτόν τον προηγούμενο Βρετανό ε, πρόεδρο της Επιτροπής μας. Ε, Και πραγματικά ευχαριστώ και του, τη συνάδελφα από την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου που ήρθε εδώ σήμερα να ακούσει τη συζήτησή μα. Είναι και αυτό ένα μέρο του προβλήματο. Γνωρίζουμε τα πρότυπα ή θα δεχόμαστε εισαγωγέ με διαφορετικά πρότυπα. Πρέπει να κοιτάξουμε να προστατεύουμε και του γεωργού ε, και κτηνοτρόφου τη Ευρώπη. Δεν μπορεί τίποτα να περνάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα παραγωγή που επιβάλλουμε στου δικού μα παραγωγού. Αυτό θα πρέπει να είναι η αρχή που να ε, διέπει την στάση τη Επιτροπή σε πολλέ από αυτέ τι πτυχέ. Δεν πιστεύονται πολλοί από του διαπραγματευτέ αυτέ τι εμπορικέ συμφωνίε εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή τέλο πάντων εκ μέρου μα ε, έλαβαν υπόψη του αυτό το στοιχείο και την δέχονται τη γραμμή αυτή. Ακούω ότι η κυρία Αγκουιλέρα το αναφέρει αυτό. Είναι μια μέρη που αφορά του πάντε, ε, όλα ένα προ ένα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε για το βόλιο, είτε για τα προϊόντα τη Ισπανία, είτε για ό,τι και αν πιάσουμε. Ε, επίσης, κύριε Κούσνοκ, να νομίζω ε, ότι ήσασταν ε, κάπως... Ε, κάπως ε, συνοπτικός τον αναφερθήκατε στο θέμα του Brexit, κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι με τις τάσεις σας και με την τοποθέτησή σα δείξατε ότι μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά αυτή είναι η δημοκρατία, αυτή ήταν η απόφαση που ελήφθηκε και η δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει να ασκείται. Ω προ την ε, θέση μα, λοιπόν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ή ακόμη και αν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μόνο του, σε κάθε περίπτωση σίγουρα οι αλλαγέ θα είναι τεράστιε για όσου μείνουν μέσα. Υποψιάζουμε, Πρόεδρε, και ελπίζω ότι θα υπάρξει μια μελέτη σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις. Ελπίζω ότι θα δούμε τι θα γίνει με τον αντίκτυπο, γιατί είναι 40 χρόνια που έχουμε εμπορικέ γεωργικέ σχέσει μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα, θα υπάρξουν τεράστιε συνέπειε για πολλού κλάδου παραγωγή, όχι μόνο στον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και εκτό. Και αυτό φαίνεται αμέσω, τουλάχιστον οι γεωργικοί κτηνοτρόφοι στην περιοχή μου, τι είπανε. Ε, τέλεια. Διότι η διακυμάνσεις στις τιμές και οι ισοτιμίες έχουν ήδη φέρει 12% αύξηση μέσα σε ένα βράδυ. Ε, ελπίζουν. Το 10% το 12% όμως που νόμιζαν ότι θα κερδίσουν από αυτό που είχαν χάσει είχε να κάνει και με άλλα πράγματα. Θα αλλάξουν οι τιμές της βενζίνης, θα αλλάξουν ε, άλλα προϊόντα και τιμές τους λόγω των ισοτιμιών. Και η αντίστροφη αλλαγή έγινε και από την άλλη πλευρά, με αύξηση 12-15% σε παραγωγούς που εισάγουν πάρα πολλά στο, προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, να είμαστε λοιπόν ε, λίγο γνώστες το τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να καταφέρουμε να τα χειριστούμε όλα αυτά. Εάν κάποιος παράγει μπορεί να αντιμετωπίσει μια αλλαγή, μια αύξηση του 2-3%. Αλλά να πάμε στο 10-15% τα όρια είναι πολύ ψηλά. Και δεν μπορεί κανείς να τα αποκριθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν άκουσα λοιπόν τις απόψεις σα. Ίσως αν θέλετε να τις ε, εξηγήσετε λίγο περισσότερο ή τέλο πάντων να μιλήσουμε μετά διμερό για όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να συμβούν και που όλοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να χειριστούμε την ερχόμενη διετία ούτω ή άλλω. Ευχαριστούμε. Τώρα λόγω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παντέρο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον καθηγητή Σουίνμπανκ για την πολύ αξιόλογη παρουσίαση και την ενδιαφέρουσα έκθεση, μελέτη. Πολύ ενημερωτική η μελέτη, ακριβής και ισορροπημένη. Όντως, οι εξωτερικές μας δράσεις και σε αυτή την κατηγορία βάζω και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, τις εμπορικές συμφωνίες, ακόμη και την COP21, τη Συμφωνία για το Περιβάλλον. Όλες αυτές οι εξωτερικές δράσεις είναι από τους σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των αγορών και διαμορφώνουν και την πολιτική και τις μελλοντικές εξελίξεις της κοινή γεωρικής πολιτικής. Αυτό που δεν έπεισε τελείως ήταν ε, η διασύνδεση που κάνατε μεταξύ των ε, μεταρρυθμίσεων του Φίσλερ και των διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ. Νομίζω ότι η μεταρρύθμιση του Φίσλερ είχε περισσότερο σχέση με εσωτερικούς ε, παράγοντες και συνθήκες παρά με τις διαπραγματεύσεις των Παγκόσμιων Οργανισμών Εμπορίου. Επίσης, δεν είναι μία μεμονωμένη εμπορική συμφωνία που έχει μεγάλο αντίκτυπο, αλλά η ισόρευση τέτοιων συμφωνιών σε συνδυασμό με την ε, αποτελμάτωση των διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ έχουμε πολύ πιο σημαντικές επιπτώσεις. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί μελέτη ε, προκειμένου να αξιολογήσει κάτι που είναι δύσκολο βέβαια, να αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο των ε, ε, διαπραγματεύσεων που τώρα διεξάγουμε και το σωρευτικό δυνητικό αποτέλεσμά τους ε, στην, και το αντίκτυπό τους στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Τώρα δρομολογούμε αυτή τη μελέτη που έχει αναγγείλει ο Αρμόδιος Επίτροπος. Ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα για να την παρουσιάσουμε και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω ασχοληθεί με θέματα οικονομικής ανάλυσης, ε, ιδιαίτερα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και θα ήθελα να σας πω ότι το βόηο κρέας ε, ήταν ανέκαθεν ένας τομέας ε, που συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή. Βρέθηκε στο επίκεντρο της ανάλυσης και της προσοχής μας και είδαμε τα μάτια μου πως διαπραγματευτέ Ένωση στις εμπορικέ διαπραγματεύσει ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί στην διαχείριση αυτού του θέματος. Και όπως είπε ο κ. Νίκολσον, πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ του υπερβολικού ανοίγματος και της, ε, ε, του πλήγματος στην Ευρωπαϊκή Γεωργία, αλλά και της ανάγκης ε, να μην χάσουμε ευκαιρίες από το άνοιγμα άλλων αγορών. Ε, βουλευτής από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου έθεσε ένα ερώτημα για τις προδιαγραφές. Το σημειώνω και την απάντηση θα την ε, αφήσω και θα την μεταβάσω στους εμπορικούς διαπραγματευτές και στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης μου, προκειμένου να σας ε, στείλουν εκείνη τις απαντήσεις. Πάντως, ε, σας διαβεβαιώ ότι οι εισαγωγές μας σήμερα πληρούν τις προδιαγραφές της ασφάλειας των προϊόντων. Τώρα, αν αποφασίσουμε στην Ευρώπη να θετήσουμε αυστηρότερες προδιαγραφές για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, αυτό είναι προς όφελος της τόνωσης της εσωτερικής ζήτησης, αλλά ταυτόχρονα και προς όφελος των ε, υπόλοιπων εταίρων μας στον κόσμο που αναζητούν πιο ποιοτικά προϊόντα. Και ως οικονομικός αναλυτής έχω διαπιστώσει την τελευταία δεκαετία διπλασιασμό των εξαγωγών των γεωρικών προϊόντων. Οπότε τα γεωρικά μας προϊόντα χαίρουν ε, ιδιαίτερης εκτίμησης ε, στο εξωτερικό και δεν είναι μύθος αυτό. Εκτιμάται ιδιαίτερη η ποιότητα των προϊόντων μας. Και από το 2008 έχουμε αυξήσει κατά πολύ τις εξαγωγές μας και έχουμε γίνει κατεξοχήν εξαγωγίας γεωργικών προϊόντων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα αθέμητο ανταγωνισμό από προϊόντα τρίτων χωρών που παράγονται με φυτοφάρμακα που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το θέμα θα το αφήσω στους ειδικού. Πάντως ξέρω ότι υπάρχουν ε, νομοθετικές διατάξεις για τα ελάχιστα κατάλοιπα σε χώρια και εισαγόμενα προϊόντα και από ό,τι ξέρω, ότι, από ξέρω οι προδιαγραφές για όλους τους ελληνικούς εμπόρους είναι ευστηρές για όλα τα προϊόντα και τα εισαγόμενα και θα πρέπει να πληρούνται ε, οι προδιαγραφές για τα φυτοφάρμακα και τις χημικές ουσίες που επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ε, ζήτησε το λόγο η κυρία Ροντρίγκε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, εμένα με ενδιαφέρει και φαντάζομαι θα προβληματίσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο του ανταγωνισμός ε, στα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τους ελέγχους των γεωρικών και μη γεωρικών προϊόντων που ε, περνάνε τα σύνορά μας. Εγώ μάλιστα είμαι σύμβουλος σε ένα ισπανικό λιμάνι και ξέρουμε τι γίνεται όταν έχουμε φρέσκα προϊόντα από την ε, Νοτιοτική Αφρική ή τη Μεσόγειο και ε, προτιμούν να μην περάσουν από το λιμάνι της Βαλένθια και να παρεκτραπούν σε άλλο λιμάνι, γιατί εμεί στη Βαλένθια εφαρμόζουμε πολύ αυστηρού ελέγχου εισαγωγή. Έτσι, υφιστάμεθα τον το ανταγωνισμό από άλλα ε, λιμάνια που έχουν πιο χαλαρέ ε, προδιαγραφές για τον έλεγχο. Αυτό σας ρώτησε. Έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό που πλήττει και τον κλάδο και την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερους κανόνες και προδιαγραφές για την ποιότητα της παραγωγής μας, αλλά θέλω να απαιτούμε, να απαιτούμε από τα εισαγόμενα προϊόντα να πληρούν τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, αλλά οι πολίτες ε, ε, αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως όργανο που φέρει συλλογική ευθύνη. Μην μας λέτε λοιπόν δεν είναι ευθύνη της δικής μας Γενικής Διεύθυνσης αλλά μιας άλλης. Θα πρέπει να είναι η συλλογική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν χρειαζόμαστε περισσότερες νομοθετικές διατάξεις αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί και αυστηροί στην υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που γίνονται να γίνονται με το ίδιο επίπεδο αυστηρότητας ε, και τις ίδιες απαιτήσει παντού. Και επίσης ε, να έχουμε τα εχέγγυα ότι όλα τα εισαγόμενα προϊόντα ελέγχονται ε, με τους ίδιους όρους και πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και προδιαγραφές με αυτές που απαιτούμε από τους Ευρωπαίους γεωργούς. Αυτά και δυστυχώς τέτοιες διαβεβαίως δεν άκουσα από την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ. Έχουμε κάποια άνεση χρόνου. Γι' αυτό και μπορώ να ξαναδώσω το λόγο και στον κύριο Χόισλινγκ. Ε, Ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπε η Κομισιόν. Είμαστε τόσο εκπληκτικός εξαγωγέας σε όλες τις διεθνείς, ε, διεθνείς αγορές και τι ωραία που είναι τα πράγματα. Εγώ όμως θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτό συνέβη μόνο λόγω της δραματικής μείωσης των τιμών των γεωργικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια. Δείτε λιγάκι τι έχει γίνει στο γάλα. Μα η τιμή του γάλακτος, ε, του ευρωπαϊκού γάλακτος είναι πλέον χαμηλότερη από εκείνο, από εκείνο της Νέας Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις επιτυχίες εντός εισαγωγικών στη Γερμανία χάσαμε τα τελευταία χρόνια χιλιάδες γαλακτοπαραγωγούς. Είναι επιτυχία αυτό. Στο χοιρινό κρέας, αντίστοιχες τάσεις. Εγώ λοιπόν αμφισβητώ το μοντέλο των εξαγωγών που έχει ακολουθηθεί. Ποιος ωφελείται εν τέλει από αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και την κατάργηση κάθε είδους προστατευτισμού. Για τις εισαγωγές και τις προδιαγραφές ε, που θα πρέπει να τηρούνται. Μα δείτε στις ΗΠΑ επιτρέπονται φυτοφάρμακα και ζυζανιοκτώνα τα οποία εμείς έχουμε απαγορεύσει εδώ και 20 χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει με δημητριακά που ήδη ε, διακινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά και τα οποία έχουν παραχθεί στις ΗΠΑ. Δεν μπορείτε να λέτε λοιπόν ότι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους. Ο κύριος Φλάναγκαν, ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν μου απάντησε η Κομισιόν ε, στο ερώτημά μου. Είναι ε, η πρώτη φορά που η παραγωγή βόηου κρέατος λαμβάνουν αντιφατικά ε, μηνύματα. Η κυρία Μάλστρομ έχει δίκιο ή ο κύριο Χόγκαν. Τελικά είναι θέμα συζήτηση και διαπραγμάτευσης στο Βόρειο Κρέα ή δεν είναι. Χρειαζόμαστε απάντηση. Και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεστε άλλος, ε, άλλωστε εδώ ε, για να μας ακούσετε και να ακούσετε τους ε, ανθρώπους που εκπροσωπούμε απαντήσατε με κάπως ασαφή τρόπο. Μπορείτε να μου δώσετε μια συγκεκριμένη απάντηση. Τι γίνεται με το βόρειο κρέας. Συζητιέται ή δεν συζητιέται. Ε, μπορεί τώρα που τελείωσε το δημοψήφισμα ο κύριος Χόγκαν ε, να έχει αρχίσει άλλο τροπάρι. Εν τέλει τι ακριβώς λέει ο άνθρωπος αυτός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματικά εκφράζω την ικανοποίησή μου που μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υπάρξει μια μελέτη για τα συνδυασμένα αποτελέσματα των διάφορων εμπορικών συμφωνιών στα εισοδήματα των Ευρωπαίων Γεωργών και κοινοτρόφων. Όμως θα προσυπογράψω και σε όσα υπόθηκαν από την σκοπιά της ανάλυσης και για τον ανταγωνισμό που δημιουργείται μεταξύ των Ευρωπαίων Γεωργών και των παραγόντων των χωρών λόγω των φυτογειονομικών μέτρων. Βεβαίω γίνονται κάποιες μελέτες για τα ζευγνιοκτώνα που περιέχονται σε εισακομμένα προϊόντα. Αυτό που, είναι, το ανέφερε και ο συνάδελφος είναι το θέμα της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαίων Γεωργών εναντί των τρίτων χωρών. Όταν σε τρίτες χώρες χρησιμοποιούνται προϊόντα που είναι απαγορευμένα στους Ευρωπαίους Γεωργούς και κάποιες φορέ με περιορισμούς από ιδιαίτερα από συγκεκριμένα κράτη-μέλη που ε, κάνουν ακόμη πιο λεπιτερό το λογαριασμό που πληρώνουν οι γεωργοί. Τελικά τι επιβάλλουμε σε αυτού του ε, Ευρωπαίους γεωργούς πότε τα εισαγόμενα προϊόντα θα σέβονται τα ίδια πρότυπα παραγωγού και όχι μόνο του προβληματισμού καταλήπων, ακόμη και αν αυτά έχουν κάποια σημασία για την υγεία των Ευρωπαϊκών καταναλωτών. Το πραγματικό πρόβλημα είναι η ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή παραγωγή. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει κάποια στιγμή απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Θα ήθελα εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να δευτερολογήσει. Παρακαλώ. Um, uh, θα προσπαθήσω να δώσω μια σαφή απάντηση στην ερώτηση που ήταν και αυτή πολύ συγκεκριμένη. Δυστυχώς, δεν ξέρω τι θα πούν και τι θα αποφασίζαν αυτή τη στιγμή ο Επίτροπος Χόγκαν ή ο Επίτροπος Μάλστρομ. Όμως, ως ερευνητής που ασχολούμαι με τα σωρευτικά αποτελέσματα αυτών των συμφωνιών και εκπονώ σχετική μελέτη, το Φεβρουάριο μου ζητήθηκε να δω τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των τελευταίων συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλους τους κλάδους, μεταξύ των οποίων για το Βόιο. Αυτή είναι η μόνη πληροφορία που έχω. Κατά τα άλλα, στα σχόλια για να τον ανταγωνισμό με προϊόντα που παράγονται με χημικά τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρώπη, θα πρέπει να το παραπέμψω στους συναδέλφους που είναι υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο ντοσχέ. Μάλιστα, αλλά παρακαλώ σημειώστε όλες αυτές τις ε, ερωτήσεις και παραπέμψτε στους αρμοδίους προκειμένου να λάβουμε γραπτός απαντήσεις. Υπάρχει και ένας άλλος ε, τομέας που είναι σχετικά έλος. Ε, υπάρχει όμως, παρόλο που είναι σχετικά αδιόρατος. Πρόκειται για την κερδοσκοπία στις παγκόσμιες αγορές. Ξέρουμε ότι οι τιμές γαλακτοκομικών προϊόντων ε, καταποντίστηκαν και τότε συνάθηκαν πολλές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης, futures, προθεσμιακές έτσι γίνονται κερδοσκοπίες ε, με βάση τις τιμές των προϊόντων. Και αυτό το είδαμε έντονα στην αγορά γάλακτος και γάλακτος σε σκόνη. Ε, συμβαίνει και στις αγορές σιτηρών, αλλά και σε άλλους κλάδους. Το θέμα της κερδοσκοπίας είναι πολύ προσεκτικό, μπορεί να είναι πιο αδιόρατο, αλλά σαφώς ε, εμφανές, παρόν μάλλον στις, στις ε, αγορές. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Γιατί η κερδοσκοπία συνιστά απειλή και για τις εθνικές πολιτικές αλλά και για την ευρωπαϊκή πολιτική, την κοινή γεωρική πολιτική. Πάντως ε, η μελέτη που αναθέσαμε στο τμήμα πολιτικών μας διαφώτισε για τις για τις αλληλεπιδράσεις των εξωτερικών δράσεων προς την κοινή πολιτική και τι ε, επιπτώσεις έχουν αυτά τα ανοίγματα των αγορών. Μερικές φορές είναι ήδη εμφανή τα αποτελέσματα αυτού του ανοίγματο. Για παράδειγμα το άνοιγμα προς τις ουκρανικές αγορές, προς τα ουκρανικά προϊόντα. Το βλέπουμε αυτό ιδιαίτερα στην Πολωνία. Αλλά δεν θα ε, περιοριστούν στην Πολωνία οι επιπτώσεις από το άνοιγμα της ε, αγοράς μας στα ουκρανικά προϊόντα, θα μεταδοθούν και προς τις υπόλοιπες χώρες, γιατί η αγορά μας είναι ενία, μην το ξεχνάμε. Θα δώσω και πάλι το λόγο στον καλεσμένο μας. Αλλά να σας υπενθυμίσω και μία συνάντηση που θα έχουμε την Επίτροπο Μάλμστρομ και τον Επίτροπο Χόγκαν τον Οκτώβριο, οπότε θα μπορέσουμε και απευθείας να τους θέσουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα ήθελα τώρα να ξαναδώσω το λόγο στον καθηγητή Σουίμπανκ για να σχολιάσει αυτή την άκουσε και να δώσει ενδεχομένω και κάποιες απαντήσεις. Παρακαλώ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έγιναν πολλές συζητήσεις. Κάποιες από αυτές αφορούσαν τα φυτογενομικά ζητήματα και τις εισαγωγές και αυτή η συζήτηση έγινε και με την ε, Κομισιόν. Ε, εγώ ε, θα ήθελα να απόσχω από αυτή τη συζήτηση γιατί δεν ασχολήθηκα με ζητήματα φυτογενομικής προστασίας. Επίσης, υπάρχουν διάφορες ε, εξελίξεις ε, που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή γεωργία, όπως είναι η διακυμάνιση των τιμών ε, και τα λοιπά, που φυσικά αξίζει να συζητηθούν. Αλλά και πάλι αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που μου ζητήθηκε να κάνω είναι να εξετάσω πώς οι εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρέασαν την γεωργική πολιτική. Ήταν πολύ σαφής ο στόχος μας. Ο κύριος Ντεκάστρο είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον να υπάρξει μια νέα έρευνα πώς η γεωργική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε και μια συζήτηση για το TTIP, για τη μερκοσούρ, για τις ποσοστώσεις ε, στο βόιο κρέας. Δεν λάβαμε απαντήσεις από την Κομισιόν ε, στα ερωτήματα του κυρίου Φλάναγκαν, αλλά από την αρχή του καλοκαιριού ε, ήταν σαφές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εξαιρεθεί το βόιο κρέας αν πρόκειται να γίνουν σοβαρές συζητήσεις με τη Μερκοσούρ. Επίσης, έχουν γίνει συζητήσεις για αυτό το θέμα, αλλά ε, η γνώμη μου είναι ότι μία εμπορική συμφωνία δεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες φυσικά και μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και νομίζω ότι οι απαντήσεις που θα περιμένουμε το φθινόπωρο θα είναι πολύ χρήσιμες από την Κομισιόν. Ο κύριος Ντέσμαντ είπε, ρώτησε... Ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία πολλαπλών ε, εμπορικών συμφωνιών ή μήπως θα έπρεπε να ανασυσταθεί ο γύρος της ε, Ντόχα. Εγώ ε, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο κάτι τέτοιο. Ένα από τα ζητήματα που ανακύπτουν από αυτές τις εμπορικές συμφωνίες είναι ο βαθμός στον οποίο εμπεριέχονται πράγματα πέραν των παραδοσιακών δασμολογικών ζητημάτων ή μέτρων ποσοστώσεων. Ένα μικρό σχόλιο ε, που συμπεριέλαβα στην έκθεσή μου είναι ε, ένα σχόλιο που έκανε ένας οικονομολόγος. Γιατί εγώ προσπάθησα να είμαι γενικά ουδέτερος ως προς το πώς οι εξωτερικές δράσεις επηρέασαν την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Είναι ένα σχόλιο το οποίο αφορούσε το πόσο έχουν ωφεληθεί οι καταναλωτές από, το, από τις εμπορικές Εγώ πιστεύω ότι αυτό ισχύει στον ένα ή στον άλλο βαθμό η ίδια η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίστηκε σε μια τελωνιακή ένωση όπου μειώθηκαν οι δεσμολογικοί φραγμοί, ε, φραγμοί και έτσι δεν ωφελήθηκαν μόνο οι παραγωγοί ε, από τα μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς αλλά και οι καταναλωτές από τις χαμηλότερες ε, τιμές και από τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων που είχαν στη διάθεση τους. Φυσικά αυτό ε, προκαλεί πιέσεις και προκλήσεις για τους παραγωγούς λόγω του ανταγωνισμού. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί με μέτρα πολιτικής. Ε, μου ζητήθηκε επίσης να συζητήσουμε το Brexit. Νομίζω ότι δεν είναι ο καταλληλότερος χώρος για να γίνει μια τέτοια συζήτηση, εδώ τουλάχιστον, αλλά με χαρά να το συζητήσουμε κάπου αλλού αν θέλετε. Εξ όσων γνωρίζω πάντως, οι Βρετανοί πανεπιστημιακοί δεν ε, έχουν ξεκινήσει ε, καμία συζήτηση για το τι πρόκειται να γίνει ε, και το ζήτημα του συνόρου με τη, στη Βόρεια Ιρλανδία είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω τουλάχιστον σε έναν βαθμό να, να απάντησα στα ζητήματα που μου τέθηκαν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Σίγουρα είναι σημαντικό να ασχολούμαστε με αυτέ τι εξωτερικέ πτυχέ και τι εξωτερικέ δράσει και το πώ επηρεάζει τη γεωργία. Ε, σίγουρα θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα γιατί έχει μεγάλες διαστάσεις και η, παγκοσμιοποίηση και η κοινή παγκόσμια γεωργική αγορά μας υποχρεώνει να λαμβάνουμε υπόψη τους εξωτερικούς παράγοντες και το πώς επηρεάζουν την ευρωπαϊκή γεωργία. Παλιά δεν είχαμε τόσο μεγάλες μεταφορές, τόσο μεγάλες αποστάσεις. Τώρα υπάρχει δυνατότητα μεταφορών σε μεγάλες αποστάσεις και έχουμε παγκόσμια αγορά. Θυμάστε όμως τι έγινε όταν ε, ε, εξεράγει το ηφαίστειο και δεν μπόρεσε να πάει η βελική σοκολάτα στην Κίνα και ε, διακόπησαν οι μεταφορές πολλών προϊόντων. Υπάρχει το πρόβλημα το συνοριακό. Ε, Επίση δεν υπάρχει μόνο το θέμα το, των πτήσεων και το κατά πώς θα φτάσει ένα προϊόν, αλλά τι γίνεται με την ασφάλεια. Θα πρέπει να προβλέπονται υψηλέ προδιαγραφέ ασφάλεια. Γι' αυτό και η εξάρτηση από την παγκόσμια αγορά έχει τα ωριά της. Και το εμπόριο είναι διμερές. Υπάρχουν δύο πλευρές. Όταν εμείς θέλουμε να ανοίξουμε την αγορά μιας ε, χώρας εταίρου και άλλη χώρα είναι λογικό να θέλει άνοιγμα και της δικής μας αγοράς προς τα δικά της προϊόντα. Είναι αμφίδρομη η κατάσταση. Και πρέπει να υπάρχει ένα δούνε και λαβήν. Και αυτό το είδαμε κατά τη μεταρρυθμίση της ε, κοινή οργάνωσης αγοράς ζάχαρης. Ε, από αυτήν ε, την μεταρρύθμιση όμως και το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς επωφελήθηκαν κυρίως οι μεγάλες εταιρείες και βιομηχανίες της Βόρειας Αμερικής και όχι η μικρή παραγωγή ζάχαρης. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά λοιπόν, πώς οι εξωτερικές δράσεις επηρεάζουν την κοινή γεωρική πολιτική. Και καλό θα είναι να επαναρχόμαστε σε αυτό το θέμα. Να ευχαριστήσω και πάλι τον καθηγητή κύριο Σουιμπάνκ, του συναδέλφους για τη συζήτηση και είχαμε κάπως την πολυτέλεια χρόνο, γι' αυτό έκανα και εγώ κάπως πιο εκτεταμένα σχέδια, σχόλια. Χαίρομαι πάντως που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την παρουσίαση αυτής της μελέτης. Το είχαμε συζητήσει και το είχαμε ζητήσει από τους συντονιστές. Χαίρομαι που επιτέλους τα καταφέραμε. Ο κύριος Φλάναγκαν, όπως είπα, έχουμε κάποια άνεση χρόνου σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, στα διάφορα και για να προχωρήσω αυτό που είπε ο κύριο Νίκολσον, το αν γίνεται να έχουμε μια έκθεση για τον Brexit ή τέλος πάντων μια ειδική συνάντηση για τον Brexit. Και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει αυτό. Είναι τεράστιο το ζήτημα για τους Βρετανούς, τους Ιρλανδούς και τεχνοτρόφους και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από την άποψη τη χρηματοδότηση και όλα τα κονδύλια που συνεισφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΚΑΤ. Θα χρειαστεί ιδιαίτερη συνεδρίαση γι' αυτό ή κάποια ακρόαση ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ καλύτερος γνώστης των μηχανισμών αυτού του σώματος, αλλά κάτι που να κάνουμε και πρέπει να γίνει. Διότι αυτή τη στιγμή συζητιέται λίγο ως ε, ζήτημα του παρασκηνίου και καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να το πούμε ευθύ αμέσω και να ετοιμαστεί έκθεση εδώ και τώρα, αλλά πρέπει να συζητηθεί. Είναι το μόνο που μας απασχολεί στην Ιρλανδία, εκτός από Εκτός από κάποια άλλα μικροζητήματα ε, που μας απασχολούν ταυτόχρονα, αλλά πραγματικά είναι το ζήτημα που απασχολεί την επικαιρότητα. Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτό. Ναι. Θα το συζητήσουμε στους συντονιστέ πρώτα. Ε, ίσως το θέσει ο κύριο Νίκολσον. Θα επανέλθουμε και θα δούμε με τι μορφή θα το διοργανώσουμε. Ωραία, ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα, ευχαριστώντας και πάλι τον καλεσμένο μας και τους συναδέλφους για τη συμμετοχή στη συζήτηση, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, ο κύριος Νίκολσον πάλι. Για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, όντως, ε, καλώς το επισημαίνει και ο συνάδελφος, αλλά έκανε και ένα σχόλιο. Πρέπει να δούμε τη δυνατότητα, γιατί όπως είπατε σωστά, και εσείς ο ίδιος πρόεδρε, τα γεγονότα είναι αυτά που είναι. Ίσως είναι λίγο γρήγορα για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Θα μπορούσαμε ίσως τους συντονιστές να δούμε πώς θα το προσεγγίσουμε. Διότι σίγουρα θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ΚΑΠ. Για όλα τα κατάλληλα. Σας ευχαριστώ. Δεκτή η πρόταση, θα το σκεφτούμε στους συντονιστές. Στα διάφορα Πρώτη και, δευτερα ε, Σεπτεμβρίου ο κύριος Στεφάν Λευκόλ, Λεφόλ, πρώην Ευρωβουλευτής και είναι Υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας, ε, είχε συνάντηση με άλλους υπουργούς ε, κρατών μελών και εκεί συζητήθηκε το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εκεί Συμμετείχε εκ μέρους της Επιτροπής Γεωργίας ο πρώτος αντιπρόεδρος μας, ο κύριος Αντριέ. Και σε επόμενη μας συνεδρίαση θα μας ενημερώσει για ε, τα αποτελέσματα αυτού του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της 1ης και 2ης Σεπτεμβρίου. Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε και για την έκβαση της διάσκεψης του CORP του ΚΟΡΚ που έγινε 5 και 6 Σεπτεμβρίου και τι συνέχεια θα δοθεί στη διακήρυξη για την ανάπτυξη πέθρου που είχε πρωτοεγκριθεί πριν από 20 χρόνια και πώς θα εφαρμοστεί με τις ε, νέες συνθήκες και την σύγχρονη πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Αυτά θα τα πούμε στο Στρασβούργο. Επόμενη συνεδρία 26 Σεπτεμβρίου. Γεια σας. Καλώς μεσημέρι.